Right. Um, Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Να σας προειδοποιήσω εκ των προτέρων ότι θα προσπαθώ να ξεκινούν οι συναντήσεις μας στην ώρα τους, χωρίς δηλαδή το ακαδημαϊκό τέταρτο της καθυστέρησης, διότι είναι άδικο όταν φτάνουμε ε, στο κομμάτι που αφορά τις εκθέσεις, ο παρουσιάζουν την έκθεσή του να αποδειχθεί ότι έχει ο λιγότερο χρόνο στη διαθέσή του. Τέλος πάντων, είμαστε στο σημείο... Α, ποιο σημείο είμαστε... Τώρα που είναι ο Hans Πίτερ Μάρτιν εδώ, μπορώ, μπορούμε να ασχοληθούμε με την απόφαση των συντονιστών. Δηλαδή, τον Ιούλιο ε, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα εφαρμόζουμε τους κανόνες του, Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου που δεν είναι ιδιαίτερη θέση στους συντονιστές στα πλαίσια της αλλά μόνο στις ομάδες και στους ε, αντιπροέδρους. Με τους νέους κανόνες Αυτή η συνάντηση είναι για τους ε, διορισμένους ε, συντονιστές. Αν δεν είστε στη ομάδα δεν μπορείτε να συμμετάσχετε. Και οι συντονιστές συμφώνησαν να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες. Ο Χάνς ε, Πέτερ Μάρτιν νομίζω είχε αντίρρηση μου είχε πει να μιλήσω δημοσία για αυτό το θέμα πάντως έχει το λόγο ο Πέτερ. Ναι, λυπάμαι που θα πρέπει να σας καθυστερήσω λίγο, αλλά μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα των βουλευτών. Εδώ έχουμε εκλεγεί όλοι επί της ίδιας βάσης και ευχαριστώ την Πρόεδρο που ακολούθησε αυτή τη διαδικασία γιατί σήμερα το πρωί δεν ήθελα να απασχολήσω τους Αμερικανούς συναδέλφους με τέτοια θέματα διαδικαστικά. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που κάνετε αυτή την επίσημη ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, μας συστήθηκε να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή για να ενημερώσω τους συναδέλφους για το τι έχει συμβεί ως τώρα. Ήταν συνηθισμένο ως ε, συντονιστές εδώ στην Επιτροπή να δίνεται και στους ανεξάρτητους ε, δυνατότητα να κατέχουν θέση συντονιστή. Αυτό κατά αναλογία και προς την εκπροσώπησή του στην διάσκεψη των Προέδρων. Δεν ε, το αντελήφθησαν οι ανεξάρτητοι, αλλά έχει αλλάξει πλέον ο κανονισμός. Θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ε, κατάργηση τους δικαιωμάτων αυτών και εγώ είμαι συντονιστή σε διάφορες επιτροπές και μου ανακοινώθηκε επίσημα ότι επί του παρόντος ε, έτσι θα έχει η κατάσταση και ελπίζω να αλλάξει αυτό. Άρα, στη βάση αυτή λοιπόν πρέπει εξ ονόματος όλων να διαμαρτυρηθώ και να σας πω ότι θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θίγονται βασικά δικαιώματα των βουλευτών οι οποίοι αντίθετα με άλλους δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αποφασιστικές προκαταρτικές συζητήσεις και γι' αυτό λοιπόν σας ε, καλώ Πρόεδρε να μας αναφέρετε τι συζητήθηκε στην συνάντηση των ε, συντονιστών, γιατί η δεν θα είναι η ίδια βάση αντιμετώπιση ε, όλων των βουλευτών. Άκουσα και φήμες ότι υπάρχουν ήδη αποφάσεις, ε, έχουν παρθεί ήδη αποφάσεις για ε, εκθέσεις και θα πρέπει να σας πω ότι επί της νομικής βάσης αυτής υπάρχει ο κίνδυνος οι εκθέσεις αυτές να μην ανταποκρίνονται στις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά με την ισότιμη δηλαδή πρόσβαση των ε, βουλευτών σε αυτές τις εκθέσεις. Εγώ προσωπικά ελπίζω να μην προκληθούν δυσκολίες και ελπίζω ότι άμεσα στην συνδιάσκεψη των Προέδρων θα βρεθεί μια λύση για το κοινό συμφέρον δηλαδή. Προκειμένου να οικοτομήσουμε μια εύρυθμα λειτουργούσε Ευρώπη. Να μην υπόκεινται τέτοιες διακρίσεις ε, οι βουλευτές. Να μην υπάρχει τέτοια ανισότιμη μεταχείριση των βουλευτών σε μια τέτοια νόμιμη, νόμιμα εκλεγμένο κοινοβούλιο. Αν ε, δεν το καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, θα απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα τεθεί προηγούμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Um, Εγώ σας ευχαριστώ. Αν ενθυμούμε καλά τη συνάντηση των συντονιστών, συμφωνήσαμε κατ' ουσία ότι θα εφαρμόσουμε τους καινούριου κανόνες. Τα πρακτικά δεν έχουν ακόμα αποσταλεί σε κανέναν. Μια ταχεία διαβούλευση είχαμε με τη γραμματεία και είπαμε ότι καλύτερα να αργήσει λίγο, να αποσταλεί το κείμενο με τα πρακτικά και να σταλεί σε όλους, παρά το αντίθετο. Α, υπάρχει και ένα λάθος από ό,τι φαίνεται που έγινε. Θα έπρεπε να έχετε λάβει τις λεπτομέρειες των διορισμών εγκαίρως, ωστόσο ώστε αν θέλατε κάτι να ζητήσετε για αυτούς να το λαμβάνατε. Τέλος πάντων, η απόφαση ελήφθη Εν το μεταξύ θα σας τηρούμε ενήμερους για το οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε προκύπτει υπό μορφή εγγράφου. Εμείς θεωρούμε ότι η ερμηνεία των κανόνων ήταν ότι οι συντονιστές μιας ομάδας έχουν κοινή θέση αλλά όχι για τους ανεξάρτητους. Μπορεί αυτό το τελευταίο να αλλάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλος συντονιστής που θέλει να σχολιάσει το ζήτημα. Πάντως θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες, ούτως ώστε η διαδικασία προσφυγής κατά τη αυτής της αποφάσεως να μπορέσει να γίνει. Θέλετε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη που σας καθυστερώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κατάλαβα σωστά. Μας δίνετε θέση σιωπηλού παρατηρητή στους συντονιστές, συγκεκριμένα σε εμένα. Σωστά κατάλαβα. Μπορώ να συμμετάχω στην συνέντευξη των ε, συντονιστών χωρίς να λαμβάνω το λόγο απάντηση της Πρόεδρου. Νομίζω ότι αυτό που εννοούσαμε είναι ότι μπορείτε να αποστείλετε ένα μέρος της γραμματείας σας. Δεν υπονοώ ότι θα πρέπει εσείς να συμμετάσχετε ως σιωπηλός παρατηρητής. Ούτε είμαι στην παρούσα φάση ε, διατεθειμένη να αναιρέσω μία απόφαση που έχουν λάβει οι συντονιστές. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανεξετάσουν οι συντονιστές, αλλά αυτό εξαρτάται από την ερμηνεία ενδεχομένως των κανονισμών. Θα προχωρήσω λοιπόν όσο πιο παρεμβατικά μπορώ, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το επιλύσει στο σύνολό του του Κοινοβουλίου, όχι προκείμενη επιτροπή και προφανώς ε, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι καλύτερα είναι να ακολουθεί μια κοινή πρακτική. Να ακολουθεί μια κοινή πρακτική, όχι να αποφασίζει ότι θέλει κάθε επιτροπή. Καλύτερα λοιπόν να υπάρξει μια γενική απόφαση. Αν σας ικανοποιεί αυτή η λύση, θα ήθελα να περάσω τώρα στο 8 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων επί των πολιτικών προτεραιοτήτων για την 7η κοινοβουλευτική περίοδο. Νομίζω ότι οι βουλευτές ε, θα έχουν λάβει το έγγραφο που έχει προετοιμάσει η Γραμματεία, το οποίο συμπεριλαμβάνει ό,τι στοιχεία έχουμε αναφορικά με το τι θα ανακύψει στην παρούσα νομοθετική περίοδο. Σκοπός της συζήτησης αυτής είναι να αξιολογήσουμε αυτά που έχουν ήδη τεθεί στη διάταξη και να πούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Αν για παράδειγμα θέλουμε κάποιες εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας ή παρόμοιες προτάσεις, μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις αυτές. Τι θα γίνει τώρα α, αφότου ολοκληρωθεί η συζήτηση. Θα συντάξω μια επιστολή προς την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών αναφορικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας, συνοψίζοντας αυτά που θα έχουμε συζητήσει. Φυσικά η επιστολή αυτή θα διαβιβαστεί και στους συντονιστές για έλεγχο της ακρίβειάς της και όταν η επιστολή λοιπόν αυτή αποσταλεί στους προέδρους ε, των επιτροπών θα περάσουμε σε μία παρουσίαση των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου. Και αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ξέρουμε ότι ο χρηματοοικονομικός κανονισμός αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Ανοίγω λοιπόν ε, τη συζήτηση και ίσως κάποια από τα θέματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε θα μας προτιμάσουν και για την ε, μετέπειτα συζήτηση που θα γίνει με τον Σιουδό Υπουργό. Γιατί τότε θα συζητηθούν ίσως τα πιο κατεπήγοντα ζητήματα. Επί αυτής της βάσης λοιπόν και στρέφομαι προς τους συντονιστές. Θέλετε κύριε Γκάουσες, να ξεκινήσετε. Έχετε σχόλια. Ή μήπως θέλετε να δώσετε το λόγο σε κάποιον άλλον πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω ότι όπως και εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση είναι πολύ σημαντικά καθώς και η συνέχεια που θα δοθεί για τις ε, νομοθεσίες που έχουν ήδη εγκριθεί Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί επίσης για τα θέματα της οικονομικής κρίσης. Σήμερα μας είπαν οι Αμερικανοί συνάδελφοι ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να αναλύσουμε τα γεγονότα. Όμως οι συμπολίτες μας είναι πλέον ανυπόμονοι. Ναι, μεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δεν πρέπει και να αργήσουμε πολύ. Αυτά από την πλευρά μου και υπενθυμίσω και πάλι ότι η ρύθμιση, η κρίση, τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης είναι βασικές προτεραιότητες και οι νομοθετικές πράξεις που έχουμε εγκρίνει είναι αποτελεσματικές και πρακτικές, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητά τους και να την ενισχύσουμε και όχι τόσο να κάνουμε νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ, κύριο Σπούλμαν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και φυσικά συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο Γκαουσές. κοιτώντα αυτά που υποβάλλατε, αυτά που υπέβαλε η γραμματεία δηλαδή, ε, σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές ε, δραστηριότητες τις οποίες είναι επικείμενες, Σίγουρα δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέα σημεία α, επικέντρωσης, νέα κέντρα βάρους. Πρέπει απλά να κοιτάξουμε αυτά που έχουμε ήδη θέσει ως προτεραιότητες. Να σας αναφέρω καταρχάς σε ό,τι αφορά την απαραίτητη νομοθετική εργασία, επειδή ακριβώς ε, ξεκινούμε μια νέα νομοθετική περίοδο και επειδή ακριβώς ε, σήμερα είχαμε και προσκεκλημένους από τη ΣΥΠΑ, θα ήθελα να τονίσω για μια φορά ακόμη το ότι πιστεύω ότι ο εξοπλισμός με τον οποίο ε, εργαζόμαστε, δηλαδή ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα, το προσωπικό και όλα τα υπόλοιπα που μας διατίθενται ως ε, βουλευτές στην Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει την ευθύνη την οποία έχουμε. Και κοιτώντας ε, και συζητώντας με τους νομοθέτες της ΕΠΑ βλέπουμε ποιες είναι οι διαφορές σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και γιατί δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ευθύνες μας και τις υποχρεώσεις μας και όποτε κυρία Πρόεδρε έχετε ε, την ευκαιρία να το τονίσετε αυτό, θα σας υποστηρίξουμε. Επίσης να τονίσω ότι χρειαζόμαστε καλή εμπειρογνωμοσύνη. Όχι μόνο εμπειρογνωμοσύνη από τους ε, λομπιίστες όμως. Δεν μπορεί να είναι εμπειρογνωμοσύνη μόνο εκείνων που πλήττονται από την νομοθεσία μας, προκειμένου να καταλήξουμε σε καλές αποφάσεις. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να τονίσω και να το σκεφτείτε παρακαλώ, είναι το εξής. Είναι φυσικά σημαντική η χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Ωστόσο, είναι σημαντικό και να κοιτάξουμε και την μακροπιστωτική διάσταση των δράσεών μας, των ενεργειών μας και να μην ξεχάσουμε την πτυχή αυτή. Όπως για παράδειγμα το follow-up του σχεδίου ανάκαμψης, προκειμένου να παρακολουθούμε στενά ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, των ε, χρηματοπιστωτικών κινήτρων που παρέχουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, ποια είναι η σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, πρωτοβουλειών και των ε, εθνικών πρωτοβουλειών των κρατών μελών. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί η Λισαβόνα 2 προκειμένου να καταρτιστεί μια ευρεία στρατηγική στην αυτή περίοδο. Αναφύρεται επίσης μια δεχόμενη έκθεση πρωτοβουλίας Μακροοικονομικά θέματα είναι ο τίτλο. Η, Λισαβόνα, η στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010 και ο ρόλος των ευρείων ε, πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών. Αυτό αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας αυτής και θα πρέπει να υπάρξει και σχετική έκθεση. Αυτό στη δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί με το Λισαβόνα 2. Θα πρέπει να υπάρξει ίσως μια ομάδα εργασίας η οποία θα είναι εγκάρσια σε όλες τις επιτροπές. Θα ήθελα να το αναφέρετε αυτό στην επίστολή σας και να δείξετε και τη σχετική ευελιξία, αν θέλετε, όταν θα το παρουσιάσετε στην διάσκεψη των Προέδρων. Uh, Ευχαριστώ. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι είχα χτες μία συζήτηση με τον Επιτρόπο Ελμούνια και θα υπάρξει μία νέα έκθεση την οποία μάλλον θα παρουσιάσει 15 Οκτωβρίου στους συντονιστές και άρα θα έχουμε κάποια νέα Σημειώνω πάντως τα όσα είπατε. Σιλβί. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Απλά πέρα από αυτή την πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη θα θέλαμε τους επόμενους μήνες να κάνουμε και ερωτήσεις στους υποψήφιους επιτρόπους να κάνουμε έναν εκ το προτέρω δημοκρατικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Um, το σημειώνουμε. Eh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εκτός από τον κατάλογο των προτάσεων αυτών υπάρχουν και άλλα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ως προτεραιότητα η Επιτροπή μας. Αποτελεσματικότητα των ε, σχεδίων υποστήριξης ε, στις επιχειρήσεις και διάσωση της οικονομίας. Για να ξεκινήσω από το πρώτο, ώστε να τον νωρίτερα και μάλλον στην Επιτροπή για τον ε, Νομισματικό Διάλογο θα πρέπει να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό τα δημόσια κονδύλια που ετέθησαν στην υπηρεσία αυτών των επιχειρήσεων είχαν θετικές συνέπειες στους ε, καταναλωτές. Δεύτερο, ποιο είναι το σχέδιο διάσωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να ανακτηθούν αυτά τα ποσά γιατί αλλιώς θα δημιουργηθεί πληθωριστική φούσκα τη στιγμή που θα περάσει η κρίση. Δεύτερο, δημοσιονομική πολιτική. Όπως ξέρουν οι συνάδελφοι, το 2005 αναθεωρήθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης όταν η Γαλλία και η Γερμανία αντιμετώπισαν προβλήματα συμμόρφωσης με το περιεχόμενο αυτού του Σύμφωνου. Το αναθεωρημένο Σύμφωνο δοκιμάστηκε και συνεχίζει να δοκιμάζεται με αυτή την κρίση. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό οι δαπάνες αυτές ε, ε, που στόχο είχαν την αναζωογόνηση της εσωτερικής ζήτησης απέδωσαν ή όχι. Διότι υπάρχει έτσι μια διάχυτη εντύπωση ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δαπανήθηκαν κονδύλια που δεν ξέρουμε που πήγαν. Σήμερα το πρωί ένα μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου είπε ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε τη φορολογία. Θα πρέπει όμως να ζητήσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα ανακτήσουμε την δημοσιονομική σταθερότητα που είναι ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο βασίζεται μια σταθερή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Επίσης η Κομισιόν δεν θα πρέπει να αγνοήσει τις ε, πολιτικές που αφορούν την Λισαβόνα 2, όπως είπε ο κύριος Μπούλμαν. Εάν θέλουμε μια πραγματική στρατηγική για την ε, ε, δεκαετία 2010-2020, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα για να δούμε αν αυτή η στρατηγική που έχουμε εγκρίνει οδηγεί στην ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. Κάτι το οποίο φάνηκε και πριν και θα φανεί και μετά την κρίση. Και εφόσον συμφωνούμε ότι οι Αμερικανοί θα βγουν πρώτα από την κρίση, πρέπει και εμείς να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Και κάτι άλλο που άκουσα σήμερα το πρωί και το αναφέρω και εδώ, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι οι μακροοικονομικές παγκόσμιες ανισορροπίες και ότι οι διαφορές μεταξύ των βασικών οικονομιών του κόσμου συνεισέφεραν, συνέβαλαν είτε στην εμφάνιση είτε στην όξυνση της κρίσης και κάτι θα πρέπει να κάνουμε από αυτού. Αντικατάσταση, γίνεται λόγος για αντικατάσταση του συστήματος Bretton Woods με κάτι διαφορετικό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί ε, και εδώ όπως και στα λοιπά διεθνή βήματα. Αυτά από την πλευρά μου σε ό,τι αφορά το έργο αυτής της Επιτροπής και σχετικά με τα όσα προτίθεται να κάνει και έχει μέχρι τώρα κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σβέν. Καταρχάς, συμφωνούμε ότι έχουμε ένα μακρύ κατάλογο πραγμάτων. Ευχαριστούμε και τη Γραμματεία για την προετοιμασία. Όντως, για πολλά θέματα μπορούμε να κάνουμε σχετική συζήτηση και να συνδέσουμε και τις εκθέσεις και τις οδηγίες. Τώρα, δύο πράγματα που θα θέλαμε εμείς να δούμε στον κατάλογο. Καταρχάς, αν δεν υπάρξει πρόταση της Κομισιόν για την κοινή ενιαία, το κοινό ενιαίο φορολογικό συντελεστή, θα θέλαμε να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε στο θέμα της εταιρικής φορολογίας. Υπάρχει μία προθεσμία για τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία επιχειρήσεων. Αν λοιπόν δεν υπάρξει πρόταση της Κομισιόν θα έπρεπε να έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας από την πλευρά μας. Επίσης θα μπορούσαμε να εξετάσουμε θέματα βοήθειας σε χώρες πέρα από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα κονδύλια που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κρίσης. Επίσης, ίσως ε, μέσω έκθεσης πρωτοβουλίας θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ποιες είναι οι συνέπειες ε, τη χρήσης δημοσίου χρήματος ε, για τις τράπεζες και, τις, και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ήταν ενδιαφέρον και επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι στιγμής ούτε έχει γίνει εκτενής αξιολόγηση ενώ έχουν δοθεί και κάποια λανθασμένα στοιχεία. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον για το κοινό αυτό. Και επίσης όσον αφορά την οδηγία για τις ε, κεφαλαιακές ε, προϋποθέσεις. Το συζητήσαμε και με τις Αμερικές και είπαμε ότι οι ορισμένες τράπεζες είναι υπερβολικά μεγάλες για να τις αφήσουμε να καταρρεύσουν αλλά και πολύ μικρές για να τις στηρίξουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κριτήρια που θα ισχύσουν προκειμένου να στηρίξουμε τράπεζες που δεν θέλουμε να καταρρεύσουν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, έχει να κάνει με την κατανομή των κονδυλίων, των δημοσίων κονδυλίων και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας κατά τη συζήτηση της οδηγίας για τις ε, κεφαλαίες προϋποθέσεις. Ναι, ναι, συγγνώμη, γιατί δυσκολεύομαι να διαβάσω τα γράμματα της γραμματείας. Όλοι Σμιτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ανησυχώ πιο πολύ για το ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στο έγγραφο αυτό, γιατί η εμπειρία μου των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η ατζέντα ήταν τόσο πλήρης που τελικά δεν ξέραμε τι να πρωτοκάνουμε. Και προγραμματίζαμε επιπλέον συναντήσεις και το καθεξής. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα της κρίσης αυτής είναι ότι δεν ξέρουμε τι πρωτοβουλία να πάρουμε τελικά. Ούτε στις ΕΠΑ ούτε στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε κάπως επιφυλακτικοί για το, όταν διατυπώνουμε το τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα, να προετοιμαζόμαστε για νέες πρωτοβουλίες. Όχι να προσπαθούμε να μπλοκάρουμε την ατζέντα για τα επόμενα δύο έτη. Αυτό πιστεύω δεν θα ήταν σκόπιμο. Θα πρέπει να αντιδράσουμε και γρήγορα και έγκαιρα όταν ανακύψουν τα ζητήματα και οι εκθέσεις. Ελπίζω το ίδιο να κάνει και η Επιτροπή βλέπουμε 20 πρωτοβουλίες ε, συναπόφασης και 11 λεπές πρωτοβουλίες. Είναι αρκετά πολύ άριθμες. Ναι, λέει η Πρόεδρος, όντως. Case um, Σας ευχαριστώ και θα πρέπει να συμφωνήσω ότι πραγματικά είναι τεράστια αυτή η ατζέντα που έχουμε ενώπιόν μας και παρά το ότι είμαι καινούρια και θέλω να μάθω, υποπτεύομαι ότι είναι πιο μεγάλη η ατζέντα από αυτή που έχουν οι άλλε επιτροπέ, Αυτό που φαίνεται να λείπει είναι κάποια στοιχεία που συζήτησαν οι βουλευτές σήμερα το πρωί, όπω για παράδειγμα η νομοθεσία για τα μπόνους. Φαίνεται να υπάρχει περιορισμένη ευελιξία για την προσθήκη θεμάτων στην ατζέντα επειδή είναι τόσο μεγάλο το εύρος της ατζέντα, αλλά θα ήθελα να ξέρω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε ε, τις διάφορες οδηγίες, όλες τους τις πτυχές που θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε περίπτωση σφαλμάτων. Να ρωτήσω λοιπόν ε, όσους ε, βρίσκονται πιο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στο Κοινοβούλιο, πώς μπορούμε να ε, εφαρμόσουμε τα λόγια που ακούσαμε σήμερα το πρωί, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι συμβαδίζουμε με την παγκόσμια νομοθεσία και πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθεί τέτοια διαιτησία όντω στη βιασύνη μας να περάσουμε αυτή την ατζέντα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίντς, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ουσιαστικά και ο Ούντο Μπούλμαν μας είπε ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι μας. Άρα είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιήσουμε εκεί που μπορούμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και άρα θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει η γραμματεία να προσπαθήσει να ελέγξει Ποιου είδους εκθέσεις, μέτρα, νομοθεστικές προτάσεις τα τελευταία χρόνια είχαν πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Γιατί το θέμα δεν είναι να παράγουμε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, αλλά να επικεντρωθούμε σε εκείνα τα προγράμματα τα οποία όντως έχουν προτεραιότητα και όπου όντως ξέρουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη πολιτική επιρροή. Τώρα αν είναι 20 πρωτοβουλίες απόφαση στις 18, ε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να διαλέξουμε τις σωστές ε, πρωτοβουλίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις πρωτοβουλίας, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά η εντύπωση που μου δόθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ότι κάναμε πάρα πολλές εκθέσεις πρωτοβουλίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μεν, αλλά στο σερτάρι κατέληξαν δε. Και με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε, πραγματικά πρέπει να αποφύγουμε τέτοια λάθη. Να μην χρησιμοποιούμε και σπαταλάμε, αν θέλετε, τους πόρους μας αυτούς ε, σε εκθέσεις που μπορεί να είναι καλές και χρυσές και άγιες, αλλά δεν έχουν επιρροή. Να δούμε πού υπάρχει πολιτική επιρροή. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερο τώρα. Το είπε και ο συνάδελφος Γκαρσία Μαγκάιο εν μέρη. Ξέρουμε σήμερα ότι η πλειονότητα των κρατών μελών έχει έλλειμμα. Γιατί ο προπολογισμό τους δεν τηρεί τα κριτήρια του Μάστριχτ. Ξέρουμε επίσης ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει φέτος, αλλά θα αρχίσει ουσιαστικά από το χρόνο και τα επόμενα χρόνια θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι το ζήτημα των κριτηρίων του Μάστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας θα τεθούν και πάλι στο προσκήνιο. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι λείπει. Θα πρέπει θεωρώ εκ των προτέρων να τοποθετηθούμε ρητά για το ποια θα είναι η αντιμετώπιση μας, γιατί θα τεθεί το θέμα αυτό και αν εκ των υστέρων τρέχουμε να το προλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε, αν το Συμβούλιο προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις, θα είναι περιορισμένη η δυνατότητα επιρροής μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συμπεριληφθεί και αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος? Αν δεν υπάρχει άλλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Α, συγγνώμη. Κυρία Γκιόρη, ευχαριστώ. Πράδρε είδα το μακροσκελέστατο αυτό κατάλογο. και δεν θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλα. Όμως υπάρχουν κάποια σημεία που δεν αναφέρονται. Τα συμπεράσματα, τα πορίσματα στα οποία καταλήγουμε από την κρίση. Δεν έχουμε μιλήσει επαρκώς για το ότι ας πούμε πολλά κρατημέλη χρειάστηκαν τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγαρία μεταξύ αυτών. Χωρίς τη βοήθεια της Ένωσης θα είχαν καταρρεύσει. Εστονία επίσης. Ρουμανία επίσης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό και κυρίως να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους κατέληξαν σε αυτήν την ε, χαλεπέστατη κατάσταση κάποια κράτη-μέλη. Τονίζει δε και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σωτήρα Θα, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα όταν συναντηθούμε τον κύριο Τρισέ. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης που δεν συμμετέχουν, που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη α, έκαναν κάποιες δηλώσεις που δεν έγιναν δεκτές α, με ενθουσιασμό. Ενώ ε, και εκδόθηκαν κάποια κρατικά ομόλογα τα οποία δεν γίνονται δεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετα, άλλα κράτη μέλη της Ένωσης που δεν είναι κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη όπως η Δανία και η Σουηδία εξέδωσαν κρατικά ομόλογα τα οποία δέχεται η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αν μη τι άλλο πρέπει να το μελετήσουμε. Τώρα, ο μακροσκελής αυτός καταλόγος αναφέρει και διάφορα θέματα που αφορούν ε, ε, φορολογικές απάτες ή φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με πορίσματα της Κομισιόν, 39,3% των φορολογικών εσόδων της ε, Ένωσης εξαφανίζονται λόγω απάτης ή φοροδιαφυγής. Είναι και αυτό ένα θέμα που θα πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω. Είναι θέμα αξιοπιστία και ευθύνη που φέρομαι έναντι των πολιτών μα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. I have Mr. Clinton. where... Where, Mr. Mr. Clinton is working, but he's coming now. There, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Um, uh, uh, um, Ο κ. ναι, θα ήθελα να αναφέρω αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ από πλευρά ε, τη ΓΚΟΕ. Η Λετωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία έλαβαν επιδοτήσει βάσει του άρθρου 119 και μα ενδιαφέρουν οι κοινωνικέ επιπτώσει τη δράση αυτής και στην πληθώρα των προτάσεων που μας ε, υποβάλατε, θα θέλαμε να προσθέσουμε και αυτή την ιδέα, είτε έκθεση πρωτοβουλίας, είτε έκθεση της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν κατά τα άλλα να υποστηρίξω και τις ε, πτυχές, τα θέματα που άπτονται της αντιμετώπισης της κρίσης. Τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο σε ό,τι αφορά την θέση των προτεραιοτήτων. I Κάτι προ διευκρίνηση. Βλέπω στα μακροοικονομικά θέματα ότι υπάρχει ετήσια έκθεση για την Ευρωζώνη, αλλά δεν αναφέρεται η ετήσια έκθεση τη ΕΚΤ, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. για, για την ίδια χρονιά. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και η αιτήσια έκθεση τη ε, ΕΚΤ. Λείπει. Θα το ξαναβάλουμε, λέει η πρόεδρος. Δεν χάθηκε. Είναι εκεί, ακόμα και αν δεν το βλέπετε. Αλλά με, με κάτι συγχωνεύτηκε, γι' αυτό δεν ε, αναφέρεται ρητά. Ο κύριος Μπούλμαν, αυτό τι σημαίνει, πρόεδρε, ότι η έκθεση της ΕΚΤ είναι κομμάτι της ε, εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας. Ναι, έχουμε την ετήσια εκθέση για το ευρώ και την ετήσια έκθεση για την ευρωζώνη. Εκεί δεν καλύπτεται έτσι και η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Right, so that, that then is missing, but it is an automatic report that... Δεν αναφέρεται λοιπόν ρητό, αλλά συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, διότι υπάρχει το πρόβλημα των πέντε εκθέσεων, ότι έχουμε δηλαδή μέγιστο βαθμό πέντε εκθέσει. Διότι αυτέ οι οποίε παγίω επανέρχονται είναι η έκθεση της ΕΚΤ κτλ. Ο κ. Μπούλμαν. Έχει δίκιο ο συνάδελφο ε, που έθεσε το θέμα η ετήσια έκθεση για την Ευρωζώνη είναι μια έκθεση για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ενώ η έκθεση της ΕΚΤ αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν ότι η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο των εκθέσεων πρωτοβουλίας. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, θα το διευκρινίσουμε. Πάντα υπάρχει ακόμα και αν δεν αναφέρεται ριστός. Είστε ήσυχος, συνάδελφε. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Μπούλμαν, σε περίπτωση που προκύψουν ανακοινώσει της Κομισιόν, όπως ας πούμε για την ε, Ευρωζώνη και για τη στρατηγική της Λισαβόνας, είναι δυνατόν να μην θεωρηθεί πρωτοβουλία η έκθεση. Έχουμε περιθώριο μία ανακοίνωση της Κομισιόν να σημάνει ότι καλούμεθα εμείς να συντάξουμε έκθεση χωρίς να ξοδέψουμε πολεμοφόδια δηλαδή από τις ε, γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίες. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έγινε στο παρελθόν. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Αλλά είναι πρόβλημα. Γιατί έχουμε ας πούμε συμφωνήσει για μία έκθεση για τον ανταγωνισμό. Υπάρχει και μια άλλη ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει ο Σονούπου Κομισιόν. Αυτά μπορούν να συνδυαστούν, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν μπορούν να συνδυαστούν. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, θα διανύμουμε έναν ε, πιο επίκαιρο κατάλογο. Ο κύριος Παντάρ Ευχαριστώ. Ακούστηκε ότι η Εσθονία ζήτησε οικονομική βοήθεια από την Ένωση για να διέλθει της κρίσης. Ουχή. Δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει. Δεν αληθεύει ε, που δεν είναι. Είχαμε επαρκή αποθέματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να αμβλύνουμε τις παρενέργειες της κρίσεως μόνοι μας. Um, Καλώς το σημείωσα. Κύριε Γκίγκολτ, σύντομα γιατί ξαναμιλήσατε. Δύο, ε, δύο σύντομα. Μια γενική κριτική των ε, εκθέσεων πρωτοβουλίας. Είναι αποτελεσματικές μόνο όταν καλούν την Κομισιόν να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Έτσι είναι, είναι αποτελεσματικές και χρήσιμες οι εκθέσεις πρωτοβουλίας. Αλλιώς όχι. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, για ε, το θέμα της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών. Συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες αυτές και όπως αποφασίσαμε στη συνάντηση των συντονιστών θα συμπεριληφθεί το θέμα αυτό και στην έκθεση για την κατάσταση της Ευρωζώνης. Ε, θα πρέπει να είναι ένα από τα σημαντικότερα φαντάζομαι ζητήματα στα πλαίσια αυτά που θα πρέπει να μελετήσουμε. Το έχουν ήδη συζητήσει και συμφωνήσει οι συντονιστές. Ευχαριστώ. Ο κ. Στόιγαν. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τα μακροοικονομικά θέματα, όπως η ετήσια έκθεση για την ζώνη ευρώ, θα ήθελα να πω ότι όλες οι χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007 δεσμεύτηκαν να αναλάβουν όλες τις δεσμεύσεις που θα τους οδηγούσαν στην υιοθέτηση του ευρώ. Οπότε η έκθεση αυτή θα έπρεπε να επικεντρωθεί μόνο στη φάση προετοιμασίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή χώρα. Ο τελευταίος ομιλητής θα είναι ο κύριος Χουάνγκο. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι επέμειναν στην μακροοικονομική θεώρηση. Είναι σωστό αυτό πρέπει να δούμε και στα πλαίσια της Λισαβόνας 2 την μακροοικονομική πολιτική. Για στη, στη Λισαβόνα 1 είτε απουσιάζει είτε δεν παρουσιάζεται με το σωστό τρόπο. Σήμερα όταν μιλάμε για πολιτική προϋπολογισμού η οικονομική πολιτική. Βλέπουμε πολλά κράτη-μέλη που θέλουν να έχουν περιθώρια ελιγμών προκειμένου να αναλάβουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και επίσης αρκετοί συνάδελφοι έχουν δίκιο που ζητούν διάλογο για το σύμφωνο σταθερότητας. Γιατί σήμερα κανείς δεν το εφαρμόσει. Βρισκόμαστε σε περίοδο ύφεσης ε, και μία πολιτική υπερβολικά περιοριστική θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην ανάπτυξη. Και βεβαίως η μείωση της ανάπτυξης θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στα φορολογικά και τελικά να οδηγήσει σε αύξηση των ελλημάτων περαιτέρω. Οπότε θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυξημένα ελλείμματα γιατί δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Ένα συνάδελφος ε, είπε επίσης ότι η κεντρική τράπεζα κατάφερε να δημιουργήσει το πρόβλημα στην Ουγγαρία Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε την αποστολή της Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα όταν έχουμε φιλόδοξα κρατικά προγράμματα βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι ίσως να μην επαρκέσουν αυτά. Σας υπενθυμίσω και το αμερικανικό παράδειγμα. Οπότε ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Κεντρική Τράπεζα να βοηθήσει τη χρηματοδότηση του δημοσίου ελλείμματος όπως έκανε και με τις ιδιωτικές τράπεζες κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Συμφωνώ με όσους είπαν ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνεται σε περιπτώσεις που βρισκόμαστε στον επιθανάτιο ρόγχο σε καταστάσεις δηλαδή όπου έχουμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με συστημικά προβλήματα όπως η Lehman Brothers όπου βεβαίως ήταν πολύ δύσκολο να διαπιστώσουμε πού ακριβώς ήταν το πρόβλημα να τσεκάρουμε τα βιβλία και να βρούμε τα προβλήματα. Και βεβαίως θα έπρεπε να αναλάβουν αυτού του είδους τους ελέγχους οι αρμόδιες ε, εποπτικές αρχές μας. Και κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μέρος μια πολιτικής σταθερότητας. Γιατί διαπιστώσαμε εν μέσω κρίσης ότι ορισμένες φορές δεν αρκεί η πολιτική ανταγωνισμού. Χρειάζεται και πολιτική σταθερότητας προκειμένου να μην ενταθεί η κρίση. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να εξετάσουμε ακριβώς τι θα έπρεπε να ενταχθεί σε αυτή την πολιτική σταθερότητας. Για παράδειγμα, Ενδεχομένως θα έπρεπε ακόμη και να απαγορευθούν ορισμένους επιθετικές εξαγορές ή συγχωνεύσεις αν διαπιστώνουμε ότι πέρα από ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική ανταγωνισμού ότι δεν υπάρχει και η κατάλληλη αντιστοιχεία διασύνδεση μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. Τώρα όσον αφορά τα συμπεράσματα για την κρίση, θα υπάρξει επιτροπή υπό την προεδρία του Βολφ Κλίντς, η οποία θα εξετάσει την κρίση, το πώς προέκυψε, τις συνέπειές της. Και επειδή η δική μας επιτροπή έχει πολλά βάρη και καθήκοντα, θα είναι χρήσιμο να έχουμε αυτή την επιτροπή Ακόμη βεβαίως δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική της εντολή, όμως σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει εμείς εδώ να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας επικοδομητικά και να μην υπάρξουν επικαλύψεις με την Ειδική Επιτροπή. Όσον αφορά τις εκθέσεις πρωτοβουλίας, όπως γνωρίζετε, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τους. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τις προφορικές ερωτήσεις και τα ψηφίσματα, που επίσης οδηγούν σε διάλογο στην Ολομέλεια. Κάτι που αυξάνει το προφίλ ενός θέματος και επίσης μας επιτρέπει να αντιδράσουμε άμεσα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε πότε θα έχουμε στη διάθεσή μας νέα έκθεση πρωτοβουλίας. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε το διάλογο με τον Jean-Claude Trichet στις 28 ε, Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να ανταλλάξουμε απόψεις και να θέσουμε ενδεχομένως και κάποια ερωτηματικά σε σχέση με το ότι γίνεται. θα συντάξουμε συμπεράσματα και θα τα διανύμουμε. Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά τους και είμαστε σχεδόν στην ώρα μας για να περάσουμε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τους ε, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Ο εισηγητής για αυτή την οδηγία είναι ο Ζαν Πολ Γκοζές. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Γκοζές για να κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε το βράδυ διορίστηκα εισηγητή Οπότε δεν μπορώ να έχω οριστική άποψη σήμερα, πολλό δε μάλλον που στην ομάδα μας α, αποφασίσαμε να κάνουμε συλλογική δουλειά συγκεντρώνοντας ε, τους ε, βουλευτές του ΕΛΚ γύρω από τον εισηγητή, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση συνενετική για ένα δύσκολο θέμα. Και λέω ότι είναι δύσκολο το θέμα, διότι όπως αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί από τους ε, ε, Αμερικάνους ομολόγους μας ότι τα hedge funds δεν φταίνε για την κρίση και ότι δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να τα ρυθμίσουμε τα hedge funds. Αυτό άκουσα από πολλούς. Α, από την άλλη είπαν πολλοί ότι τα hedge funds έχουν ύποπτο ρόλο, στρεβλωτικό ρόλο, διότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτά με στόχο άμεση κερδοφορία, χωρίς να σκέφτονται δηλαδή στο το απότερο ε, μέλλον μακροεπενδυτικά, μακροοικονομικά αν θέλετε. Με όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνολική θεώρηση της κατάστασης. Πολλά είναι τα προσυζήτηση σημεία. Το πρώτο είναι εάν περιοριζόμαστε σε αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Δηλαδή δυνατότητα α, διορισμού managers για τα επενδυτικά αυτά ταμεία ή αν το πάμε πιο μακριά, ευρωπαϊκό διαβατήριο που όπως προτείνει η Κομισιόν μετά από τρία χρόνια θα μας ε, δώσει τη δυνατότητα να θέσουμε στο εμπόριο ε, και μη ευρωπαϊκά προϊόντα. Το θέμα αν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια επί της χρήσεως αυτών των ε, hedge funds. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να μελετήσουμε, να αξιολογήσουμε και να αναπτύξουμε και βεβαίως είναι καλοδοχούμενοι όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να μου γνωστοποιήσουν τη θέση τους για να την λάβω υπόψη μου. Ούτως ώστε να μην είναι αγαπητέ Ουνο οι ε, αυτοί που θα αποφασίζουν για το περιεχόμενο των εκθεσεών μας αλλά οι ευρωβουλευτές. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ετοιματή του συνάντησα τον δήμαρχο του Λονδίνου σήμερα που ερχόταν με αντιπροσωπεία από το City την οικονομική δηλαδή καρδιά του Λονδίνου για να συζητήσουμε τα hedge funds και εγώ δήμαρχος είμαι με 309 ψυχές έχει βέβαια η κοινότητα ε, της οποίας είμαι δήμαρχος ενώ αυτός είναι ε, δήμαρχος του Λονδίνου ιδιαίτερα συμπαθής με άκρος ικανοποιητικά γαλλικά ηρίστο εμπαρόδο. Έτσι τον δέχτηκα και έτσι ε, ε, θεωρώ γενικά τα πράγματα και οι συνάδελφοι που ήταν παρόντε και την τελευταία θητεία γνωρίζουν ότι αυτά τα πράγματα γίνονται διότι οι δύο βασικέ εκθέσει που είχα την δυνατότητα να παρουσιάσω ε, για τι υπηρεσίε πληρωμέ και για τι ε, ελέγχου εγκρίθηκαν με ευρία πλειοψηφία και μπορέσαμε με την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι εγκρίνουμε σε πρώτη ανάγνωση. Κάτι το οποίο καταδεικνύει και τη βούλησή μα να τοποκριθούμε ε, γρήγορα και αποτελεσματικά στα καυτά επίκαιρα ερωτήματα. Η νομοθεσία εξάλλου ε, από τη φύση της πλέον στις μέρες μας ε, δεν χαράσεται στο μάρμαρο, δεν ισχύει για 100 χρόνια. Μέρα με τη μέρα μπορεί να αλλάξει. Ε, αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι στο ρυθμό των αλλαγών. Αυτά. Ε, και θα συνεργαστώ με τους Σκιώδης, ε, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία για το άκρος αυτό τεχνικό ζήτημα. Η προπαρασκευαστική αυτή δουλειά είναι απολύτως απαραίτητη. Ευχαριστώ. Thank you. I will take... Σας ευχαριστώ να ακούσουμε τον κύριο Μπούλμαν γιατί δεν έχουμε σκιώδη από την ομάδα σας. Άρα προφανώς είσαστε εσείς υπεύθυνος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο τον εισηγητή. για την πολύ χιουμοριστική του προσέγγιση σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαι αφελής βέβαια και ξέρω ότι ο οικονομικός κόσμος έχει συμφέροντα και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξουμε ποτέ. Απλά απευθύνω έκκληση προκειμένου η γνώση μας, η εμπρογνωμοσύνη μας, η ικανότητά μας και η ευφυΐα μας ε, με την οποία προτείνουμε καλή νομοθεσία να είναι αντίστοιχη και να συμβαδίζει με την ευφυγία εκείνων αυτών που έχουν ήδη την νομοθεσία αυτή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους ε, εκείνους στο Κοινοβούλιο που υπέδειξαν στον ε, εισηγητή Ράσμουσεν και στον εισηγητή Λένε ότι ως νομοθέτες σήμερα είμαστε στην ημερήσια διάταξη και ότι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση και ότι αυτά που είπε ο συνάδελφος Κίγκολ προκειμένου οι σωστές εκθέσεις πρωτοβουλίες να έχουν επιρροή και να καταλήξουν σε νομοθεσία αυτό θα γίνει μόνο αν αναγκάσουμε τους, ε, τα θεσμικά όργανα να δραστηριοποιηθούν επιτέλους και θα πρέπει λοιπόν αυτό να το διατεπιστώσουμε και να το συνειδητοποιήσουμε και στην Επιτροπή αυτή. Όταν λάβαμε αυτή την πρόταση πριν από τον ε, προεκλογικό αγώνα, το θέμα ήταν να ρυθμιστούν οι managers. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το εξής. Καταρχάς, θα θέλαμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία ζημιάς στην Ευρώπη. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον ρόλο των hedge funds και να ρυθμίσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο και αυτό στα πλαίσια μιας σύγχρονης νομοθεσίας. Κατά δεύτερον, φυσικά και έχουμε συμφέρον να ρυθμιστούν τα προϊόντα αυτά τα οποία διατίθενται στην Ευρώπη προκειμένου να έχουν υψηλή ποιότητα, υψηλό επίπεδο. Να είμαστε, αν θέλετε, το επίπεδο σύγκρισης και να θέσουμε και κρίσιμα ερωτήματα και να κάνουμε και κριτική. Να ρωτήσουμε αν η αδιαφάνεια, το βραχυπρόθεσμο αυτή η ομίχλη, αν θέλετε, που σχετίζεται με τους ε, παράγοντες αυτούς, διευκρινίζεται στα πλαίσια της πρότασης της Επιτροπής. Θα πρέπει να αποφύγουμε να ανοίξουν καινούργια κενά. Και επίσης, ε, μήπως ε, με μία ανεπαρκή νομοθεσία όντως επιτρέπουμε σε τρίτες χώρες να είναι ανταγωνιστικές προς τις δικές μας. Να κοιτάξουμε τους οικονομικού μας τομείς και να δούμε μήπως όντως μειονεκτούν οι τράπεζές μας. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να ειδωθούν και στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο πύχης στις συζητήσεις μας. Θέλουμε καλύτερη ρύθμιση και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Εννοείται, εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί σε περίπτωση που ο κλάδος, οι ενώσει καταναλωτών μας επιστήσουν την προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα. Μας πούνε ότι κοιτάξτε υπάρχουν συνέπειες ε, τις οποίες δεν έχετε εξετάσει, για παράδειγμα, εμπειρικές συνέπειες ε, μιας ενδεχόμενης νομοθεσίας και χρειάζεται διάλογος. Ε, αυτό είναι αυτονόητο. Thank you. Um, next on... Σας ευχαριστώ. Επόμενος ε, στον κατάλογο ο κύριος, η κυρία Στήλερ. Η Κάθριν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται μια τέτοια πρώτη συζήτηση και χαίρομαι που το βάλαμε στις τέσσερις, γιατί αλλιώς μπορεί να μην προφταίναμε κιόλα. Αλλά νομίζω ότι ο ανοιχτό χαρακτήρας που το ανοιχτό πνεύμα που επιδεικνύει ο εισηγητής είναι πολύ θετικός και πολλοί με έχουν ήδη προσεγγίσει για την νομοθεσία αυτή. Είναι λοιπόν εξαιρετικά κρίσιμο, εξετάζοντας το θέμα αυτό, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες προκειμένου να κάνουμε διαφορά και να αλλάξουμε τους κανόνες για να είναι αποδοτικές. Ο Ούντο μίλησε για τα κενά. Αυτό είναι ένα από τους μεγάλους φόβους ότι αν δεν, τα κάνουμε, αν δεν κάνουμε καλή ρύθμιση θα δημιουργήσουμε πιο πολλά προβλήματα. Στη Σκοτία, την οποία και εκπροσωπώ, επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τα private equities. Μίλησε και ο συγκριτής και για αυτά και για τα hedge funds. Αυτό περιλαμβάνει και άλλα επενδυτικά μέσα, κάποια εκ των οποίων φαίνεται ότι εμπλέκονται χωρίς να ευθύνονται. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, οι επενδυτικές εταιρείες που καλύπτονται από την νομοθεσία αυτή, ενώ ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν υπεύθυνε για την οικονομική κρίση. Και καλύπτονται από πολλές ευρωπαϊκές νομοθεσίες, άρα θα πρέπει να σκεφτούμε σωστά αν θα μπορούσαμε να έχουμε μία ένδειξη του χρονοδιαγράμματος που έχουμε μπροστά μας, γιατί φυσικά ε, ο χρόνος πιέζει. Και είπε και ένας συνάδελφος ε, από τους φιλελεύθερους ότι αυτό απασχολεί και την Επιτροπή. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει το νομοθέτημα αυτό να έχει τον ανάλογο χρόνο που του αντιστοιχεί. Να μην τον περάσουμε βιαστικά, που επιδεικνύει τέτοιο ανοιχτό πνεύμα ο εισήγητης και είμαι βέβαιη ότι πρόκειται να ακολουθήσουν και πολλέ συζητήσει και τι επόμενε εβδομάδε, του επόμενου μήνε. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Κάνφιν. Je suppose Μάλλον εμένα εννοούσατε. Είμαι ο ισκιώδης ε, εισηγητής των Πρασίνων για αυτή την οδηγία. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με τον κύριο Κοζέσα. Χαιρόμαστε που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με αυτού του είδους τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου εδώ και αρκετά χρόνια ακούμε επικρίσεις για τα κεφάλαια αυτά και για τους συστημικούς κινδύνους που δημιουργούν για όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είχε συζητηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1990 και πλέον είμαστε καθυστερημένοι στην αντίδρασή μας αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. αυτή είναι η υπεύθυνη της κρίσης. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει συνένεση για αυτό. Και κυρίως όχι τόσο η απουσία νομοθεσίας, αλλά το πώς παρακάμφθηκε αυτή η νομοθεσία. Οπότε σήμερα, αν θέλουμε να έχουμε μία συνεκτική πολιτική, η οποία θα δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη και τα μακροοικονομικά στοιχεία, πρέπει να εξετάσουμε και αυτό το θέμα γιατί τα hedge funds ακόμη και αν δεν αποτέλεσαν το βασικό λόγο της κρίσης ήταν ένα από τα εργαλεία της. Επίσης, είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τα κεφάλαια υψηλού κινδύνου, γιατί είναι από τα πιο επικίνδυνα εργαλεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό εξάλλου είναι και τα πιο αποδοτικά. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ρύθμιση νομοθεσία για το πιο επικίνδυνο κομμάτι του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και θα ήθελα να κάνω εδώ ένα παραλληλισμό με την βιομηχανία την απλή. Συνήθως εκεί ασχολούνται ακόμη περισσότερο με τα πιο επικίνδυνα εργαλεία. Θα έπρεπε λοιπόν το ίδιο να γίνει και εδώ με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι παρόλο που έχουμε αυτή την πολύ επικίνδυνη δραστηριότητα, δεν είχαμε ζητήσει καμία ασφάλιση για τους ιοδιωτικούς αυτούς οργανισμούς. Ο μόνος δηλαδή που ασφάλιζε τα hedge funds είναι ο ίδιος ο φορολογούμενος. Κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα κάθε εταιρεία να ασφαλίζεται για το κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σε άλλους. Όπως ακριβώς γίνεται για την ασφάλιση αυτοκινήτου. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ασφάλιση προκειμένου το κόστος της ασφάλισης να το αναλάβουν πράγματι αυτοί οι ιδιώτες. και θα πρέπει να υπάρχει και μεγάλη κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται σήμερα από την οδηγία. Και όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο τους διαχειριστές αλλά τα ίδια αυτά τα κεφάλαια είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και πρέπει να επαναξετάσουμε στην οδηγία. Τέλος. Δεν θα έπρεπε εδώ να θεω κάποιοι οποίοι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εταιριών και κάποιοι που είναι κατά των εταιριών. Εγώ γνωρίζω και πολλές εταιρείες, ειδικά μικρομεσαίες, οι οποίες υποφέρουν εξαιτίας της ε, κατάστασης σήμερα, οι οποίες υποφέρουν εξαιτίας ε, των όσων έγιναν με τα hedge funds. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με υπεράσπιση κάποιων εταιρικών συμφερόντων, αλλά με υπεράσπιση των συμφερόντων καταρχάς του φορολογούμενου πολίτη και κατά δεύτερο λόγο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Uh, Ευχαριστώ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Καμάλ και μετά στον κύριο Κλίντς. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω και ως σκιώδης εισηγητής της συντηρητικής ομάδας. Θα συνεργαστούμε, ελπίζω, επικοδομητικά με τον εισηγητή και επί της οδηγίας αυτής. Εγώ ως εκπρόσωπος του Λονδίνου Προφανώς θα έπρεπε να ενδιαφερθώ για την πρότασή σας. Και είναι αλήθεια ότι μας ανησυχεί το θέμα της περιορισμένης ανάπτυξης του τομέα στο Λονδίνο και στην Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των hedge funds βασίζονται στο Λονδίνο. Ενδιαφέρει λοιπόν συγκεκριμένα τους δικούς μου ψηφοφόρους το θέμα. Όμως ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο. Και σίγουρα και εμείς στο Λονδίνο ενδιαφερόμαστε να δείξουμε ότι διδαχθήκαμε από την κρίση και ότι θα οδηγηθούμε σε μια νομοθεσία χωρίς παραθυράκια. Γι' αυτό επικροτώ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν προκάλεξαν την κρίση τα hedge funds. Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι και να κατανοήσουμε επίσης και τις διαφορές μεταξύ hedge funds, equity κτλ. Είναι αλήθεια ότι τα hedge funds έχουν ε, πολλά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια που επενδύονται με κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά έχουμε το private equity που έχει πιο μακροπρόθεσμες βλέψεις. Να πω και κάτι άλλο. Συχνά υπάρχει μία φιλική, ένας φιλικός ανταγωνισμός μεταξύ Λονδίνου και άλλων οικονομικών κέντρων όπως το Παρίσι για παράδειγμα. Δεν πρέπει όμως να το δούμε έτσι το θέμα. Θυμηθείτε ότι στη Σαγκάη, στο Τόκιο, στο Ντελαουέρ όλοι προσπαθούν να προσελκύσουν αυτοί τις οικονομικές δυνάμεις και αδειμονούν. Τέλος, όποιες και είναι οι απόψεις σας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είτε θεωρείτε ότι αποτελεί πληγή για την κοινωνία, είτε κάτι πολύ χρήσιμο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποια θα είναι η επίδραση στους ψηφοφόρους μας. Και η αλήθεια είναι ότι με φοβίζουν κάποιες συνέπειες της αρχικής οδηγίας για τις ιδιωτικές ασφάλειες, κάτι που ενδιαφέρει πολλούς από εμάς, ειδικά το θέμα των ιδιωτικών συντάξεων. Εγώ, συζητώντας ε, με εργαζόμενους ε, της ε, περιοχής μου, που εργάζονταν σε μια εταιρεία η οποία εξαγοράστηκε. Αυτό που μου είπαν ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε τα συνταξιοδοτικά ταμεία αυτών των ανθρώπων και ότι δεν πρέπει να τους περιορίσουμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ταμεία. Επίσης, δεν πρέπει πάντα να έχουμε ως μοναδική δυνατότητα της τα δημόσια ταμεία, γιατί έχουμε πολλές επιχειρήσεις που πλέον, ακόμη και ταχυδρομικές και άλλες επιχειρήσεις που πλέον βρίσκονται σε συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και θα χρειαστούν αυτού του είδους τα ταμεία, τα ιδιωτικά. Πέρα από αυτά όμως, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες, τις αρνητικές συνέπειες, ειδικά αυτές που δεν ήταν ηθαλιμένες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τι είναι το κατάλληλο να κάνουμε για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι η Επιτροπή μας υπέβαλε τόσο γρήγορα μία πρόταση σε ό,τι αφορά τις ε, εναλλακτικέ επενδύσεις και σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές. Αλλά επέλεξαν ένα θέμα. Εγώ είμαι από τη Φρακφούρτη, έχω από το Λονδίνο. Και θα μπορούσα να με ενδιαφέρει ε, να περιοριστούν οι δραστηριότητε στο Λονδίνο, αλλά συμφωνώ με τον συνάδελφο Καμάλ. Ο κίνδυνο είναι να μην φύγουν οι επιχειρήσει και να έρθουν ε, από το Λονδίνο στο, στη Φραγκφούρτη, αλλά να πάνε στην Ελβετία ή οπουδήποτε αλλού. Και χαίρομαι που ο Βρετανό συνάδελφος συντηρητικό αποκαλύπτει ότι είναι πραγματικά μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιθυμεί να παραμείνει. Δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα αυτά και πραγματικά χαίρομαι που ε, το διαπιστώνω αυτό. Καταρχάς, αντίθετα με διάφορους που εξέφρασαν την, ε, το θαυμασμό του για την πρόταση αυτή, εγώ πρέπει να πω ότι η δική μου άποψη ενδιαφέρει. Μου φαίνεται ότι προσπαθούμε με μία οδηγία, με ένα κανονισμό, δεν ξέρω καν τι θα προκύψει τελικά, να ρυθμίσουμε ταμεία τα οποία είναι τόσο διαφορετικά, μάλλον πόρους που είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους στη σύνθεσή τους και στην ουσία τους. Είπαμε ότι θα πρέπει να διακρίνουμε τι είναι το hedge funds, τα private equities και ούτε καν τα hedge funds δεν είναι όλα ίδια μεταξύ τους και συγκρίσιμα. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι η προσέγγιση αυτή την οποία ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή One Size Fits All ένα για όλα δηλαδή, είναι πολύ προβληματική. Νομίζω ότι με την προσέγγιση αυτή δεν πρόκειται να πετύχουμε το στόχο μας και σίγουρα όταν προσπαθούμε με έναν κανονισμό να διεκπαιρεώσουμε ολόκληρο το θέμα αυτό, θα πρέπει να προβλέψουμε διαφορετικές, μεμονωμένες ε, νομοθεσίες για τα διάφορα αυτά εργαλεία και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει ε, επί του τελικού αποτελέσματος το Δεκέμβριο, είναι υπερβολικά φελαιόδειξο. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Τώρα. Πρόκειται για μία πρόταση η οποία είναι εξαιρετικά αντιφατική και θα πρέπει μέσα από τις συζητήσεις μας να επιλύσουμε αυτές τις αντιφάσεις. Κατά δεύτερον, προστατεύεται με αυτή την πρόταση ένας κύκλος ατόμων ο οποίος ενδεχομένως να μην χρειάζεται να προστατευτεί γιατί πρόκειται ίσως για θεσμικούς επενδυτές και όχι για τον ε, χύψη καθημερινό πολίτη. Αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές θα έπρεπε να ξέρουν και ξέρουν συνήθως με τι ασχολούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες κατηγορίες, θα πρέπει να πω το εξής. Τα private equities, τα οποία δαιμονοποιούνται ιδιαίτερα στη χώρα μου και τα hedge funds. Κοιτώντας ε, αντικειμενικά τα στατιστικά στοιχεία, πέρα από τις μεγάλες και πολλές αποτυχίες, δεν το αμφισβητώ αυτό, παντού υπάρχουν, τελικά όμως πιο πολλέ θέσει εργασία δημιουργήθηκαν και σώθηκαν παρά καταστράφηκαν. Άρα από πλευρά δημοσιοοικονομική η, η συνεισφορά του, η συμβολή του. Γι' αυτό λοιπόν προειδοποιώ να αντιμετωπίσουμε και να εξετάσουμε αυτό το θέμα, αλλά να μην εικάζουμε ότι πρόκειται για εργαλεία τα οποία πρέπει να τα περιορίσουμε και να τα ελέγξουμε πλήρως. Όχι. Δεν σημαίνει φυσικά αυτό ότι δεν πρέπει να αναπτύξουμε σχετική νομοθεσία. Σίγουρα. Αλλά να έχουμε και ένα μέτρο. Να προσέξουμε κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τη λύση των τρίτων χωρών. Να μην περιορίσουμε την ροή, την εισρωή κεφαλαίων προς την Ευρώπη, όταν δεν υπάρχει ανάγκη φυσικά. Να μην δηλαδή αυτό σαμποσταριστούμε. Σε ό,τι αφορά τις ε, αποθηματικές τράπεζες. Να περιμένουμε μέχρι ότου λάβουμε τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε. Σε οκτώ εβδομάδες θα τις έχουμε τις προτάσεις αυτές, κάτι τέτοιο. Γιατί? Θα είναι μεγαλύτερες οι θεσμικές επιδράσεις στην περίπτωση αυτή. Και αυτό θεωρώ είναι προβληματικό σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή από το πάνω από 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει επίσης να το συζητήσουμε. Αν είναι σκόπιμο να γίνει αυτή η διάκριση ή μήπως καλύτερα να πούμε ότι δεν υπάρχουν όρια. Και επίσης δεν είναι σαφές πώς η μήπω καλυτερα να πουμε οτι δεν υπαρχουν ορια και ιδουγία θα ενταχθεί στο ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιμο. Έχουμε διάφορες οδηγίες για διαφάνεια και το καθεξής. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να συμβαδίζουν το ένα με το άλλο. Γιατί κοιτάξτε, ήδη ο κόσμος είναι απέραντα περίπλοκος και κάθε οδηγία, κάθε κανονισμό που εκδίδουμε περιπλέκεται περαιτέρω. Αν τώρα σε ένα τέτοιο ετερογενή τομέα όπως ε, οι εναλλακτικές επενδύσεις προκαλέσουμε μεγαλύτερο βαθμό περιπλοκότητας, αυτό ουσιαστικά θα έρθει και θα επιδεινώσει, θα κάνει σχεδόν αδύνατη τη μελλοντική λειτουργία της οικονομικής ζωής και θα συνεπάγεται μεγαλύτερη γραφειοκρατία και κόστος, χωρίς να έχουμε πετύχει ουσιαστικά τίποτα. Τελευταίο στοιχείο που θέλω να θέξω. Καταλαβαίνω βέβαια την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη διαφάνεια και για μεγαλύτερη πληροφόρηση. Ωστόσο, να προσέξουμε. Μήπως τελικά με τη ρύθμιση ενός τμήματος ε, των μέσων αυτών τελικά καταλήξουμε σε μία ε, ανισομέρεια, ανισότητα. Αν ζητάμε δηλαδή ε, πληροφορίες από κάποια συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, στρατηγικές πληροφορίες, ίσως προκληθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δηλαδή, ε, κάνω κάτι για τις εταιρείε αυτές, το οποίο δεν απαιτώ από τις κανονικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα, να προσέξουμε για να πετύχουμε κάτι θετικό, πληροφόρηση και ενημέρωση των εργαζόμενων, αλλά Μήπω από την άλλη τελικά καταλήξουμε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω ποια είναι η πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αντιτίθεμαι. Αλλά θεωρώ ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα τελικά το οποίο ε, θα μας ωφελεί όλους στο σύνολό μας συνυπολογίζοντας τα πλανεκτήματα, τα μειονεκτήματα, το κόστος, ούτε καθεξής. Αυτό θα είναι δύσκολο έργο. Εγώ ως εισηγητής για τους φελευθέρους είμαι έτοιμος να συνεισφέρω. Αλλά σας το λέω από τώρα δεν πρόκειται να είναι εύκολο το έργο αυτό. Um, Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να λάβει μέρος σε αυτή τη συζήτηση, θα σας πω ποιους έχω σημειώσει, την κυρία Λούλινγκ, την κυρία Σίρμπινγκ, την κυρία Ντατή, την κυρία Φόρντ, την κυρία Πινγκ και εγώ. Και μετά, αν λοιπόν δεν υπάρχει άλλο, θα δώσω σε αυτού το λόγο, μετά στην Κομισιόν και μετά στον εισηγητή. Να κλείσω τον κατάλογο. Ωραία. Άστριντ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Γκοζές, όταν είπε στην εισαγωγή του ότι πρόκειται για ένα δύσκολο και επίμαχο ζήτημα δεν θα μπορούσε να πει μεγαλύτερη αλήθεια. Εκ πείρας όμως γνωρίζω ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά δύσκολους φακέλους σαν και αυτόν λόγω της ε, αμεροληψίας του αλλά και της ε, εμπειρογνωμοσύνης του. Λοιπόν, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες των θεμάτων που θα συζητήσουμε και σε άλλες συνεδριάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για κάποιες αρχές. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μην νομοθετήσουμε σωστά. Ίσως ό,τι αφορά το γιατί αυτής της πρότασης. Εξού ορμάται αυτή η πρόταση. Τα hedge funds, όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν ορισμένοι, δεν είναι υπεύθυνα για την ε, δημοσιονομική κρίση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα τιμωρήσουμε εντό εισαγωγικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την απόφαση να προτείνει να τα πλαισιώσει λόγω του συστημικού κινδύνου που εγκυμονούν και όχι λόγω της ε, λάθος λειτουργίας τους. Είναι νομίζω σημαντικό να το τονίσουμε. Ε, κατόπιν, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Είναι πολύ πιθανό αυτά τα hedge funds να τα βάλουμε στο πλαίσιο κάποιων συγκεκριμένων κανόνων, αλλά θα πρέπει όποτε αυτό είναι δυνατό, όποτε αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει λέγω η νέα αυτή νομοθεσία να είναι συνεπής και να συνάδει με αυτά που ήδη υπάρχουν. Ας πούμε, οδηγία έκα και άλλα. Και προσοχή, δεν θα πρέπει να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, διότι ο κίνδυνος θα ήταν να οικοδομήσουμε ε, ένα σύστημα κατακερματισμένο όπου οι πρωταγωνιστές, οι επενδυτές, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πελαγώσουν. θα τα χάσουν. Εγώ ένα κομμάτι των διακοπών μου το αφιέρωσα μελετώντας αυτή την πολύ επίμαχη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύπλοκη, αντιπαραγωγική θα έλεγα και νομίζω ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί επί πολλών μετόπων και στοιχείων για να καταστεί αποτελεσματική. Τέλος να πω ότι θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε κάποιες βασικές αρχές που αποτέλεσαν λόγους ε, των μέχρι τούδε επιτυχιών μας σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση του οικονομικού χώρου. Και για να χρησιμοποιήσω έναν εφημισμό, ε, εκπλήσωμαι όταν διαβάζω ότι ορισμένες ε, χώρες προτείνουν ε, προϊόντα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό των συνόρων τους να υπόκεινται μόνο σε εθνικούς κανόνες και οι ευρωπαϊκοί κανόνες να αφορούν μόνο τα διεθνή προϊόντα. Αυτό ειλικρινά σας λέω με κάνει να ανατριχιάζω. Θα σημάνει το θάνατο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να απορρίψουμε με όλες μας τις δυνάμεις τέτοιου είδους προτάσεις. Διότι αλλιώς τι κάνουμε εδώ. Ας κατεβάσουμε τα ρολά και ας πάμε να πουλήσουμε στραγάλια. Κάτι τώρα πιο γενικό. Η μεταχείριση των τρίτων χωρών. Απευθύνω έκκληση να εξευρεθεί ισορροπημένη λύση σύμφωνα με αυτά που κάναμε και μέχρι τώρα. Η Ευρώπη δεν είναι μπάτε σκύλοι λέστε και αλεστικά μη δώσετε, αλλά δεν είναι και ερμητικά κλειστό οχυρό. Και από αυτού σύμφωνο πλήρως με τον κύριο Κλίντς θα πρέπει να εξευρεθεί μια λύση που να οδηγήσει σε μια ισότιμη βάση για όλους με σωστή παρακολούθηση και έλεγχο. Συμβιβασμός, μέση λύση, χρυσή τομή χρειάζεται. Αυτά για μένα είναι ορισμένα θέματα που αφορούν αυτό που αρχικά ονόμασα βασικές αρχές που διέπουν τα της λειτουργίας μας. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε ο κύριος Λίντσεν που μίλησε πριν από μένα κυρίως με αυτό που είπε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον καιρό να οριμάσει όπως έλεγε ο Φρονσουά Πάντως πιστεύω ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθεί επί πολλών σημείων και να γίνουν βαθιές τομές. Και εγώ θα συνεργαστώ με τις ταπεινέμους δυνάμεις με τον εισηγητή για να το επιτύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Κέιτ Σουίμπερν. Ευχαριστώ. πολύ πιο εύγλωτα από ό,τι θα τα έλεγα εγώ. Είπαν οι συνάδελφοι πολλά που θα ήθελα να πω. Εγώ θα περιοριστώ σε ένα διδικαστικό σημείο. Για ουσιαστικές και ως εκ τούτου σημαντικές ε, οδηγίες ε, παρουσιάζεται συνήθως και μία ε, μελέτη αντικτύπου οικονομικής φύσεως αλλά για αυτή την οδηγία δεν υπάρχει έγγραφο που να καταδεικνύει τις ε, δημοσιονομικές συνέπειες της πλήρους εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Και το λέω αυτό διότι για τα συνταγματικά ταμεία, ε, για τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και τις επιδόσεις ε, των κρατών μελών δεν έχει γίνει καμία εκτίμηση. Τι λέω? Λέω ότι αν είναι πολύ πολύ πλοκό να κάνουμε μελέτη αντικτύπου γιατί κάνουμε αυτή την νομοθετική πράξη. Γιατί υποβάλλει αυτή την νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μας μπορεί να ζητήσει τη δική της μελέτη αντικτύπου για μια συγκεκριμένη οδηγία. Αυτό το γνωρίζω. Ε, αν η Κομισιόν λοιπόν δεν μπόρεσε να το κάνει, μήπως θα έπρεπε Μήπως είναι, είναι δυνατόν να το κάνουμε εμείς, να παραγγείλουμε δηλαδή μια τέτοιου είδους μελέτη αντικτύπου. θα απαντήσει φαντάζομαι η Κομισιόν. Η κυρία Ντατή. Euh, Ευχαριστώ. Ε, ναι, και εγώ συμφωνώ γενικά με όλες τις παρατηρήσεις των συναδέρφων, ακόμα και των πρασίνων, ακόμα και των φιλελευθέρων. Παρ' όλα αυτά, να υπενθυμίσουμε ότι δημοσιονομική κρίση είναι η δημοσιονομική κρίση που έχει μετά συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Το είπε και ο κύριος Κλίντς. Αλλά όχι απορρίθμιση, όχι πλήρης απουσία ε, κανόνων. Διότι εκεί ε, ε, οφείλεται η αποτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Τα hedge funds πρέπει να είναι πιο διαφανή. Αυτό αποτελεί επιταγή και παρόλο που συμφωνώ ότι δεν είναι τα μόνα τουλάχιστον υπεύθυνα για την κρίση, θα πρέπει να τα πλαισιώσουμε σε πολύ πιο διαφανή βάση και βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε τον κατακριματισμό που ανέφερε κάποιος συνάδελφος των προϊόντων της ή των, της αγοράς και να έχουμε μια σφαιρική γενικότερη θεώρηση του οικονομικού συστήματος για να αποφύγουμε και άλλες κρίσεις στο μέλλον. Έχω επίσης επιφυλάξεις το σχέδιο οδηγίας επί του ότι τα μία τρίτων χωρών μπορεί να έχουν ε, διαβατήριο για τρία χρόνια, ευρωπαϊκό διαβατήριο για τρία χρόνια. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε βεβαίως ε, τα μία ή προϊόντα τρίτων χωρών τέλος πάντων να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Αλλά όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Και το λέω αυτό διότι αν εγκρίνουμε, αν δώσουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο σε, τρίτα, σε προϊόντα τρίτων ε, χωρών, ε, θα φτάνουν προϊόντα offshore ε, στην Ένωση και θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα όπως με τους φορολογικούς παραδείσους. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, μια αντικειμενική αξιολόγηση ε, των μέτρων αυτών. Ένας, ε, αναφέρεται ένας ανεξάρτητος αξιολογητής. Αυτό δεν υπάρχει στη Γαλλία. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο, ε, ένα τρόπο που να, είναι, που να μπορεί να ισχύει, να εφαρμοστεί για όλους. Ευχαριστώ. Η Βίκη Φόρντ. Ευχαριστώ πολύ. Με ανησυχεί πολύ η σύγχυση που φαίνεται ότι διακατέχει διάφορους ομιλητές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Τι είναι hedge fund, τι είναι private equity και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να κατανοήσουμε τις ενδυνάμει συνέπειες κάποιων διατάξεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ στην περιοχή μου έχω το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, έτσι, θα το έχετε ακούσει όλοι. Και ως ε, αποτέλεσμα της αριστείας ε, του ε, Πανεπιστημίου πολλές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που συνεργάζονται και με άλλα πανεπιστήμια έρχονται στο Cambridge για να καινοτομήσουν γιατί αυτό το χρειαζόμαστε για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις βασίζονται σε private equities, σε ιδιωτικά δηλαδή ταμεία που τους παρέχουν τους οικονομικούς πόρους για να κάνουν τη δουλειά τους μία μικρή ρήτρα σε αυτό το κείμενο που σημαίνει ότι μια επιχείρηση θα πρέπει να δίδει περισσότερα στοιχεία ε, να τα δημοσιεύει πολλά περισσότερα από ότι μια τράπεζα σημαίνει ότι μπορεί αυτές οι επιχειρήσεις να μην επενδύουν στην Ευρώπη αλλά να πάνε στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Κίνα εκεί όπου δεν υπάρχει τόσος έλεγχος και τέτοια αυστηρότης. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις συνέπειες αυτών των μέτρων. Για τα hedge funds. Δεν είναι όλες οι επενδύσεις επί των ε, hedge funds επικίνδυνες. Υπάρχει ένα ταμείο που, ε, hedge fund δηλαδή, το οποίο επενδύει σε κρατικά μόνο ομόλογα γερμανικά, ολλανδικά και γαλλικά νομίζω. Οπότε θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Αυτό το έγγραφο, όσο έχει συνταχθεί, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τι σημαίνει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υποστηρίζω πλήρως την εκπόνηση μιας μελέτης αντικτύπου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έπινγκ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένη ότι, πεπισμένος ότι έχετε πολλές ερωτήσεις για την ε, οδηγία αυτή και για κάθε νομοθεσία και κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτείται μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του οικονομικού τομέα και της ελεύθερης κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Διάβασα την οδηγία αυτή στις διακοπές και εργάστηκα επί πέντε χρόνια στην κυβέρνηση του κ. Μπόλκονσταν στην ε, Γενική Διεύθυνση, αν θέλετε, εμπορίου και με αυτή την ε, εμπειρία διάβασα την οδηγία αυτή. Υπάρχει λοιπόν ε, στην οδηγία αυτή μία διάσταση που είναι κατά της αγοράς και βλέπουμε με μεγάλη σαφήνεια ότι αρχικά, αρχικά υπήρξε ένα lex specialis για τα hedge funds, το οποίο και τροποποιήθηκε στη τελευταία στιγμή πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Τροποποιήθηκε σε lex generalis για να συμπεριληφθούν και τα venture capitals και τα private equities. Είναι λοιπόν ίσως θέμα πολιτικής και πολιτικής ε, υπερβολικής δραστηριοποίησης αν θέλετε, ίσως η Επιτροπή να άργησε να ξυπνήσει και συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα και προέβη σε υπερβολικές ε, δράσεις ε, μικροδιαχείρισης. Να σας επιστήσω την προσοχή στην διάρθρωση της οδηγίας αυτής. Υπάρχουν 7-8 σημεία όπου αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα λάβει εφαρμοστικά μέτρα, implementing measures. Δεν είναι τα πλέον απλά στοιχεία αυτά της οδηγίας. Επίσης διατυπώνεται ως η μόχλευση και η equivalence, η ισοτιμία. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να μας εξηγήσει όλα αυτά και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μείνει πίσω γιατί η Επιτροπή θα συνεχίσει, θα προβεί σε επιτροπολογία και τελικά θα προκύψει η νομοθεσία. Το equivalence τώρα, το οποίο συζητήσαμε και σήμερα το πρωί, θα πρέπει να υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ των όσων ρυθμίζονται στην Ευρώπη και στην, ε, στη ΣΥΠΑ. δεν θα υπάρχουν καινοτομίε, δεν θα υπάρχει κεφάλαιο κινδύνου, η οικονομία θα μετακατασταθεί στις ΙΠΑ. Ε, Βλέπουμε λοιπόν τις ε, συνέπειες Μάλλον βλέπουμε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αξιολογήσει ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη ύπαρξης συμβατότητας μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Τελικά θα καταλήξει από οικονομικής άποψης η Ευρώπη ένα τεράστιο γυροκομείο, αν δεν υπάρχουν τα κεφάλαια αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το κεφάλαιο που αφορά το equivalence θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Θα πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προτιμούσα να είχε μείνει στην αντίληψη του Επιτρόπου Μακρύβη η Επιτροπή, δηλαδή στο Lex Specialis, όχι στο Lex Generalis, το οποίο δυστυχώ αντιμετωπίζουμε σήμερα. Um, Ευχαριστώ. Θα περιοριστώ σε ορισμένα ελάσσονα σημεία και μετά θα αναφερθώ σε κάποια διαδικαστικά πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή και στον εισηγητή, γιατί νομίζω ότι είναι σχετικά και τα διαδικαστικά. Καταρχά, όσον αφορά την επικάλυψη με άλλες οδηγίες, για παράδειγμα τη MIFID πέρα από την οδηγία που ανέφερε και ο κύριος ε, Κλίνς, καθώς και την έκθεση Rasmussen, κοιτάξτε, ναι, θέλουμε να καλύψουμε τα πάντα, αλλά όχι να τα δίπλο ή τρίπλο καλύψουμε. Όταν μιλάμε για κίνδυνο, πρέπει να μας ενδιαφέρει και το ποιος είναι ο επενδυτής. Είναι θεσμικός επενδυτής ή άτομο, λιανική επένδυση δηλαδή. αν συζητάμε το θέμα αναπροϊόν, αυτό θα μας δυσκολεύσει στις, ε, για τους επαγγελματικούς χρήστες και τα επαγγελματικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλύτερο να προσπαθούμε να βρούμε πρακτικές λύσεις και όχι να περάσουμε σε μία εξέταση αναπροϊόν. Επίσης, εδώ θα ήθελα να δω ποιοι είναι αυτοί που χάνουν στο τέλος. Γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε πιο πρόσφατα στοιχεία για τις συνέπειες στα συνταξιοδοτικά ταμεία των απλών ανθρώπων. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία βεβαίως δεν επενδύουν όλα τα χρήματά τους σε hedge funds, αλλά θέλουν να έχουν και κάποιες τέτοιου είδους επενδύσεις με μεγάλη απόδοση, προκειμένου να μπορούν να δώσουν καλές συντάξεις όταν χρειαστεί. Επίσης με ανησυχεί η προσέγγιση της τρίτης χώρας καθώς και η προσέγγιση που προτείνεται για τις εγγύσεις στα αποθεματικά. Και επίσης τίθεται και το θέμα της Αφρικής που μένει ανοιχτό και θυμηθείτε ότι υπάρχουν και πολλές ηθικές ανησυχίες εδώ και ηθικές επενδύσεις που θα ήθελαν να δουν πολλοί από εμάς. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι η ανάπτυξη στην Αφρική είναι εξίσου σημαντική με τα hedge funds. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Τώρα, ετέθησαν ερωτήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε με τον εισηγητή. Δεν ξέρω αν γνωρίζει το πότε θα είναι έτοιμη η έκθεση. Πάντως, αν θέλουμε να μπορούμε να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης στις 9 Νοεμβρίου για παράδειγμα, τότε θα πρέπει να είναι έτοιμο το σχέδιο έκθεσης μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για να γίνουν στη συνέχεια οι μεταφράσεις. Αυτό είναι το πιο γρήγορο χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τώρα, να πω ότι υπάρχει η εκ των προτέρων αντίληψη ότι θα προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε μεταξύ μας. Και το αναφέρω απλά ως διαδικαστικό. Πάντως δεν θα έπρεπε να μειώσουμε τον χρόνο που θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Πολύ ωραία λοιπόν αν θα έχουμε έτοιμη τη θέση του Συμβουλίου μέχρι τα Χριστούγεννα, όμως εμείς από την πλευρά μας θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς είμαστε ένας δημοκρατικά ελεγχόμενος οργανισμός και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και δεν θέλουμε κάτι τόσο σημαντικό να περάσει γρήγορα και κλεισμένων το θυρών. Δεν θέλουμε να αποκλειστούν μέλη από την συζήτηση. Βλέπω αρκετούς από εσά να γνέφουν καταφατικά. Γνωρίζουν τι συμβαίνει και από την προηγούμενη θητεία ορισμένη. Αυτά λοιπόν επί των διαδικαστικών. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής. Και είναι αλήθεια ότι μας πιέζει πλέον ο χρόνος, οπότε θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. και μετά θα δώσω το λόγο και στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος ακριβώς όπως μου το ζητήσατε. Να πω καταρχάς ότι χαίρομαι για την ατμόσφαιρα στην πρώτη συνεδρίαση και χάρηκα που άκουσα και τα γενικά σχόλια που συμφωνούν με τους βασικούς στόχους της πρότασής μας. Επίσης, ε, χαίρομαι για το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θέλετε να ακολουθήσετε, παρόλο που δεν είναι ακόμη οριστικό. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σας πω ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να συζητήσουμε αυτό το θέμα ανοιχτά και επικοδομητικά. Όπως είπατε και εσείς, αλλά και ο εισηγητής. Και ανοιχτοί θα είμαστε και στις σχέσεις μας με το Συμβούλιο Ήδη εδώ και κάποιες εβδομάδες έγινε μία πρώτη πιο λεπτομερή συζήτηση επί του θέματος και με το Συμβούλιο λοιπόν θα συνεργαστούμε ανοιχτά και επικοδομητικά προσπαθώντας να παίξουμε το ρόλο μας ως διασμεσολαβητές. Τώρα, συγκεκριμένα για αυτά τα μέσα ανέφεραν οι περισσότεροι τους στόχους μας με αυτή την οδηγία. Να πω ότι οι στόχοι αυτοί, οικονομική σταθερότητα, προστασία από τους συστημικούς κινδύνους, η διάσταση της εσωτερικής αγοράς που προσπαθούμε να εισάγουμε σε αυτό το τομέα και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, προστασία του καταναλωτή. Όλα αυτά είναι πολιτική στόχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να βελτιωθεί από τη συζήτηση εδώ. Εμείς γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ρόλος μας, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία πρόταση η οποία θα είναι καλή, αναλογική, επαρκής για την επίλυση των προβλημάτων. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας. Ένα τελευταίο σημείο, ίσως πιο πολιτικό αυτή η πρόταση δεν προσπαθεί να ευνοήσει κάποιες επενδύσεις σε σχέση με άλλες, να ευνοήσει ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν σε σχέση με άλλο. Δεν υπάρχει πρόθεση τιμωρίας κανενός. Απλά θέλω να έχουμε ένα πλαίσιο ρυθμιστικό πιο επαρκές πιο διαφανές που θα βασίζεται σε ορισμένα θέματα σημαντικά για εμάς γιατί τελικά αυτό που θέλουμε είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αυτό είναι προς συμφέρον όλων, καταναλωτών, πολιτών, επενδυτών όπως ακριβώς είχατε επικέσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοζέσα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις παρεμβάσεις. Όπως είπε και η Άστριτ, σίγουρα θα έχουμε πολλές τροπολογίες, 800, 900, κάτι τέτοιο μπορείτε να περιμένετε. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Όμως, χρειάζεται και συζήτηση και αυτή την ανάγκη συζήτησης θα πρέπει να τη συμβιβάσουμε με τις φιλοδοξίες μας για το χρονοδιάγραμμα. Προκειμένου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στα τέλη αυτού του έτους ή στις αρχές του επόμενου μου φαίνεται πολύ φιλόδοξο θα πρέπει να δούμε τις διαπραγματεύσεις με την Προεδρία και την Κομισιόν βεβαίως όσον αφορά το θέμα της συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση και πολύ συχνά οι συζητήσεις στο Συμβούλιο κρατούν πολύ περισσότερο από ό,τι εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό πάντως που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανακοινώσουμε την δεύτερη συζήτηση επί του θέματος. Εγώ θα προσπαθήσω να προετοιμάσω την έκθεση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω. Συμφωνώ να προσπαθήσουμε για συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Συμφωνώ να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όμως θα πρέπει να έχουμε και λογικές προθεσμίες και βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία και με τους χειώδεις εισηγητές και με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ευχαριστώ. 6 Οκτωβρίου η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα θα βγω λίγο έξω για να υποδεχθώ τους Σουηδούς Υπουργούς. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση που είχαμε. Um, Παρακαλώ. Ησυχία. Λάβετε θέσεις για να συζητήσουμε το σημείο 9 της ημερησία διατάξεως ανταλλαγή απόψεων με τους Σουηδούς Υπουργούς. Θα ακούσουμε πρώτα τον Άντερ Μπόργκ ασκώντα την Προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ μόλις ολοκληρώθηκε μια άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ θα μας ε, μιλήσει ε, για ε, θέματα αρμοδιότητός του μετά θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό των Περιφερειακών Αγορών και μετά στα μέλη της Επιτροπής στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε στη θέση μας κυρία Μπόργκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για μας που είμαστε εδώ σήμερα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Προεδρίας μας και να ακούσουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας και βεβαίως να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις που θα θέλετε να μας ε, θέσετε. Είναι προφανές ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ένωσης σε μια πολύ κέρια καμπή της οικονομικής τουλάχιστον ιστορία μας, μας λόγω της κρίσεως βεβαίως. Η αντιμετώπιση της οποίας είναι η βασικότερη πρόκλησή μας. Μια άλλη προτεραιότητα είναι βεβαίως οι κλιματικές αλλαγές όπου θέλουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση πριν την Κομπενχάγη. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις ε, που αναφέρονται στην πραγματική οικονομία. Πέντε είναι οι βασικές μας προτεραιότητες. Ε, η βελτίωση της εποπτείας της μουσουλμικής αγοράς, ο επανακαθορισμός υγιών δημοσίων οικονομικών, η αντιμετώπιση της αγοράς απασχόλησης, ε, η αναζωγόνηση της Λισαβόνας μετά το 2010 και ε, όθηση στις διαπραγματεύσεις ε, για το κλίμα. Για την εποπτεία. Υπάρχει νομίζω ευρεία συμφωνία σε όλα τα κράτη-μέλη ότι ένα κομμάτι του προβλήματος που μας οδήγησε σε αυτή την οικονομική κρίση ήταν έλλειψη κανονιστικού πλαισίου, ε, έλλειψη ελέγχου ε, επί των τραπεζών που γίνονται διεθνείς ενώ τα νομισματικά και οικονομικά μας θεσμικά μέσα όχι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι διαρθρώσεις, οι δομές στις οποίες βασιζόμαστε να ε, εδράζονται σε μια κοινή πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μακροοικονομικά θέματα όπου ελήφθη μια πολύ καλή απόφαση τον Ιούνιο στο ΕΚΟΦΗΝ και που ευλογήθηκε αργότερα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ε, χαιρετίζουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν που θα παρουσιάσει 23 Σεπτεμβρίου. Να τονίσω το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πεποίθησή μου ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επί του θέματος για να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια του ε, φετινού φθινοπόρου. Οι κεφαλαϊκέ απαιτήσει για τις τράπεζες θα πρέπει να αυξηθούν, θα πρέπει να μειωθεί η προκυκλικότητα. Εν ώψη της ε, συνάντησης ε, της ομάδας των 20 είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για τα υπερβολικά μπόνους. Οι αμοιβέ ε, των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων είναι σαφές ότι αποτελούν κομμάτι του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Επίσης, σαφές είναι ότι αν θέλουμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα, ε, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος, να θέσουμε ένα τέλος σε αυτήν την ε, τακτική των πόνου και των αποζημιώσεων. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την όξυνση της ε, ανεργίας και να κάνουμε κάποιες διαστατικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας. Από την ε, σημερινή μας ε, συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ καταλήξαμε σε μια ε, ισχυρή νομίζω ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα προωθήσουμε στο Λονδίνο και το Πίτσπορ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη που λάβαμε την Κομισιόν, το έλλειμμα κατά μέσο όρο θα είναι της τάξης του 7% του ΑΕΠ το 2010. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό η επόμενη πρόβλεψη να αναθεωρηθεί. Ελπίζω να αναθεωρηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε αυτό, διότι είναι πολύ πιθανό να επιδενωθούν ακόμα περισσότερο τα, δημοσιονομικά των, ε, τα δημόσια οικονομικά των κρατών ε, μελών. Μάκρο πρόθεσμα, τα δημόσια οικονομικά των ε, κρατών μελών δεν ε, είναι βιώσιμα ο πληθυσμός γυράσκει υπάρχουν πολλές δαπάνες ε, λόγω των συνδεξιωτικών συστημάτων συστημάτων πρόνοιας του συστήματος υγείας όλα αυτά συντελούν στη μη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών εφόσον υπάρχουν τέτοια θέματα μακροπρόθεσμα και εφόσον υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα χρειάζεται μια διέξοδος μια στρατηγική διεξόδου. Εμεί χαιρετίζουμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει τι συζητήσει αυτέ στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ που θα λάβει η χώρα στι αρχέ Οκτωβρίου, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε τι σχετικέ συζητήσει, διότι είναι σαφέ είναι σαφές, λέγω, ότι η οικονομική πολιτική με την ευρία έννοια θα πρέπει να είναι ε, ουσιαστική ε, και να περιλαμβάνει ως δυνατόν περισσότερα θέματα. Και αυτό το λέω διότι ε, δεν αξιοποιούμε το δυναμικό που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται επεκτατικές πολιτικές. Δηλαδή, αν θέλουμε να εξαγοράσουμε ελαστικότητα, θα πρέπει βράχη και μέσω πρόθεσμα να είμαστε αξιόπιστοι. Δηλαδή, θα πρέπει να εργαστούμε εντός του συμφώνου είναι θέμα αξιοπιστία αν θέλουμε να επαναφέρουμε αυτού στην τάξη. Οι εκθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου θα δημοσιευθούν. Θέλουμε βεβαίω να δούμε τι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική εξόδου. Αλλά βλέπουμε και τι εκθέσει για την ε, μακροπρόθεσμη αηφορία που θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο των συζητήσεων στο ΕΚΟΦΗΝ κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Να υπογραμμίσω και το εξή η αξιοπιστία της του μακροπρόθεσμου πλαισίου μας για την φορολογική πολιτική είναι απαραίτητη αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ελαστικότητα, flexibility. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την μεταχείριση που θα στο θέμα της στρατηγικής αυτής. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Είναι προβληματική η κατάσταση σε πολλές χώρες, η απασχόληση μειώνεται, η ενεργεία αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να μελετούμε και θέματα αγοράς εργασίας. Η πολιτική απασχόλησης και η πολιτική ενέργεια είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής, δημοσιονομικής κρίσης και η αποφυγή της συρρήκνωσης της ζήτησης. Αλλά η δεύτερη και τρίτη γραμμή άμυνας είναι η ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, ενεργής ε, δράσης ε, για την απασχόληση ε, και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας και βεβαίως και άλλες σχετικές πολιτικές που θα βελτιώσουν την ελαστικότητα και την λειτουργία της αγοράς απασχόλησης. Αυτό είναι σημαντικό θέμα συζήτηση για την Σουηδική Προεδρία. Τώρα, ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Ε, θα συνεργαστούμε στενά ε, με την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία επ' αυτού του θέματος. Νομίζω ότι είναι σαφείς οι αρχές επί των οποίων βασιζόμαστε για να βελτιώσουμε την μακροπρόθεσμη μεγέθυνση στην Ευρώπη. Μετά της εφαρμογής των νομοθεσιών μπορούμε να κάνουμε πρόοδο. Θέλουμε όμως να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα του Προεδρείου εν ώψη του... της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Βεβαίω, και είναι στο προσκήνιο το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Χθε λάβαμε ε, τη νέα έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών από το Λονδίνο. Οι αλλαγέ ε, είναι τόσο ε, οξύε και τόσο σοβαρές που θα πρέπει κατά πάσα να αντιληφθούμε να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα. Εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ισχυρά συμπεράσματα στο ΕΚΟΦΗΝ για τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές τον ε, Οκτώβριο, στις 20 Οκτωβρίου. Και βεβαίως θα έχουμε συζήτηση και για τις κλιματικές αλλαγές, για τη χρηματοδότηση του περιβάλλοντος και την φορολογία της ενέργειας στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ. Όλα αυτά είναι κομμάτι των προπαρασκευαστικών έργων εν ώψη της Κοπενχάγης. Όπως επίσης είπα, εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε στενά στο ΕΚΟΦΗΝ ε, ε, μεταξύ των κρατών μελών για ε, όρου αναφορά για όλη την ε, Ευρώπη στα πλαίσια τη συνάντηση τη ομάδα των 20. Από την άτυπη σημερινή μα συνάντηση νομίζω ότι έχουμε ήδη κάνει πρόοδο από αυτή τη αγούση για πολλά από τα ζωτικά σημεία οι μηχανισμοί, τα μπόνου, η χρηματοδότηση του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Υπάρχει μια σαφή ευρωπαϊκή θέση πλέον, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να κινήσουμε τα πράγματα προ την κατεύθυνση που θέλουμε ε, μετά το Pittsburgh. Στον φορολογικό τομέα. Και εδώ βεβαίω ε, πολλά πρέπει να κάνουμε. Καταπολέμηση της απάτης, ηλεκτρονική τιμολόγηση στα συστήματα ΦΠΑ και βεβαίω η ε, αιτήσια έκθεση του 2010 που θα πρέπει να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδριασής μας εγκρίθηκε τον Ιούλιο το σχέδιο για το 2010 θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε ικανοποιητική λύση για, στο κοφήν του Νοεμβρίου. Μιλώ για τον προπολισμό του 2010 Αυτά εκ μέρου μου. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εκ νέου για τη δυνατότητα που μα δίνετε σήμερα να είμαστε εδώ και δίδω το λόγο στον συνάδελφό μου. Yes, please continue. Thank you. Ναι, συνεχίστε αν θέλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ τους φίλους από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες, αν θέλετε, αναφορικά με τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις σχετικές υπηρεσίες. Να σας αναφέρω ότι η Σουηδική Προεδρία σκοπεύει να αποτελέσει έναν εντερό με τον οποίο θα συνεργαστείτε και ο οποίος θα σας ακούσει προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές κρίσεις οι οποίες θα πλέξουν τους πολίτες μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν στενά και είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάει η συνεργασία μας εδώ σήμερα. Ξέρω ότι η Επιτροπή αυτή εδώ και καιρό έχει ενδιαφερθεί για τα θέματα αυτά και συνεργάζεται επικοδομητικά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει την ποιότητα των νομοθετικών πρωτοβουλειών και την ταχύτητα της έγκρισης τους. Και πολλές φορές μάλιστα σε πρώτη ανάγνωση, από ό,τι βλέπω. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ένα βασικό καθήκον για τη Σουηδική Προεδρία θα είναι να αντιμετωπίσει τις ε, ρυθμιστικές αδυναμίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις οποίες αποκάλυψε η κρίση. Και γι' αυτό λοιπόν βελτιώνουμε την εποπτεία στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ξεκινάμε λοιπόν, μιλώντα για την εποπτεία, από την αφετηρία ότι όλοι συμφωνούμε πλέον να ότι υπάρχει ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το τρέχον σύστημα για να αποτραπούν μελλοντικέ κρίσει και για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή και του επενδυτή. Έχουμε μία εντολή από το Συμβούλιο του Ιουνίου προς αυτή την κατεύθυνση και αν υπομονούμε να λάβουμε τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εργασίες στη σχετική ομάδα του Συμβουλίου θα ξεκινήσουν από τη στιγμή που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι σχετικές προτάσεις στις 23 Σεπτεμβρίου. Και επίσης προετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο είναι πολύ βαρυφορτωμένο. Τον Οκτώβριο θα απαντήσουμε εκ μέρους του Συμβουλίου αναφορικά με την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί ως τότε και είμαι βέβαιος ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα συνεργαστούν με επικοδομητικό τρόπο για να διασφαλίσουν την γρήγορη έγκριση του κρίσιμου αυτού νομοθετικού πακέτου, χωρίς φυσικά αυτό να θέσει εν κινδύνο την ποιότητα του περιεχομένου του. Και ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ μαζί σας για αυτήν την πραγματικά καινοτομική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των διαφόρων τομέων των χρηματοπιστωτικών αγορών. Νομίζω ότι αυτή η κρίση κατέστησε σαφές ότι η υφιστάμενη νομοθεσία έχει κάποια κενά. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος εδώ, αλλά υπάρχει Γενική Παγκόσμια Συμφωνία ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει για τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε κανόνες για τα ιδρύματα και για τα προϊόντα τα οποία επί του παρόντος δεν ρυθμίζονται. Το ξέρω. Ξέρω ότι συζητήσατε τα hedge funds πριν από την συνάντηση αυτή και θα έχετε φαντάζομαι ερωτήσεις. Θα χαρώ να τις ακούσω και θα πρέπει να τοποθούμε ε, σε ό,τι αφορά τις ε, επισφαλείς, αν θέλετε, ε, πρακτικές αναφορικά με τις αμοιβέ. Τώρα, να περάσω σε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με τις προτάσεις αυτές. Καταρχάς, οι σημαντικές νομοθετικές προτάσεις για τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τράπεζες, σε ό,τι αφορά την οδηγία δηλαδή συγκεκριμένα για τις κεφαλαιοκές ε, απαιτήσει. Η πρόταση του Ιουλίου δημιουργεί κανόνε προκειμένου οι τράπεζες να έχουν καλές πρακτικές αναφορικά με τις αμοιβέ και αλλαγές για τις δραστηριότητες της ε, εμπορικές των συναλλαγών και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για περίπλοκα ε, προϊόντα. Τον Οκτώβριο η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για να γίνουν και άλλες αλλαγές στην τραπεζικό κόσμο και να εισαχθούν κανόνες που επιτρέπουν στις τράπεζες να δημιουργήσουν, αν θέλετε, αποθεώματα ε, αντικυκλικά. Σκοπεύουμε λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτά τα σημαντικά θέματα και φυσικά ανυπομονούμε και στον τομέα αυτό να συνεργαστούμε μαζί σας. Κατά δεύτερον, μία οδηγία για τους ε, διαχειριστές των εναλλακτικών επενδυτικών μέσων. Πρόκειται για μία από τις ε, προτεραιότητες που ορίστηκε από το G20 να επεκταθεί δηλαδή η φυστάμενη νομοθεσία σε όλους τους παράγοντες, σε όλες τις ενέργειες οι οποίες συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, τη χρυσή τομή σε ό,τι αφορά την εποπτεία των hedge funds και των άλλων επενδυτικών εργαλείων για να κλείσω λοιπόν την παρουσίαση αυτή. Η Σιωτική Προεδρία πιστεύει ότι είναι πραγματικά κρίσιμο να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών, βελτιώνοντας την ενσωμάτωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, εγγυούμενη φυσικά και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και τον ανταγωνισμό. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια νομοθεσία η οποία θα λειτουργεί εύρυθμα με υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω άλλη μια φορά ότι αν να συνεργαστώ με εσάς, με την Επιτροπή σας, για να πετύχουμε την μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη, που πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητοι οι πολίτες μας, θέλουν πραγματικά και περιμένουν από εμά να αντιδράσουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Um, um, ευχαριστώ. Εκ μέρους του ΕΛΚ Ποιος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ ε, αγαπητοί Υπουργοί. Είχα τη δυνατότητα να συζητώ και με τους δυο σας ε, πριν το καλοκαίρι όπου εξετάσαμε τον κατάλογο των προτεραιοτήτων της Σουηδικής ε, Προεδρίας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πριν την επίσκεψή σας είχαμε σήμερα το πρωί μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της Αμερικανικής ε, Γερουσίας μάλλον του Αμερικανικού Κογκρέσου. και ενημερώσαμε αλλήλους για το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Είναι προφανές ότι η πρώτη προτεραιότητα ε, είναι η δική σας αρμοδιότητα, δηλαδή της Σουηδικής Προεδρίας. Γι' αυτό επιτρέψατε μου, αγαπητοί συνάδελφοι που τα έχετε ξανακούσει, να επαναλάβω ορισμένα σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε κάποια τακτικά αλλά και έκτακτα μέτρα για τη ρευστότητα. Η ανησυχία αυτή τη Επιτροπή του Κοινοβουλίου είναι να γνωρίζουμε μέχρι ποιο βαθμό αυτά τα μέτρα ρευστότητα για τι τράπεζε ε, φτάνουν την σωστή χρονική στιγμή και αν ναι τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε αυτά τα μέτρα που ξοδεύουν δημόσιο χρήμα. Δεύτερο, εγκρίθηκαν έκτακτα μέτρα, εξαιρετικά μέτρα για τη διατήρηση της ρευστότητος. Αγορά δηλαδή ενεργητικών των τραπεζών, κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει και από μια στρατηγική διεξόδου, εξόδου στο μέλλον. Θα ήθελα και από αυτό τη γνώμη σας. Ο Υπουργός Οικονομικών και η οικονομία έχει τεράστια ευθύνη στο θέμα αυτό για το σύμφωνο σταθερότητος ομιλό που γίνεται σεβαστό ε, τους ε, καιρούς των παχιών αγελάδων και το οποίο κανένας δεν σέβεται όταν έχουμε κρίση. Το 2005 έπληξε μικρές χώρες, αργότερα μεγάλες η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ε, το ενέκρινε αυτό μια γενική αμνηστία ούτως είπε, μια χαλάρωση των κανόνων του συμφώνου ε, στην ουσία σύμφωνο δεν υπάρχει πλέον ένας Αμερικάνος ε, βουλευτής είπε ότι δεν μπορεί να εξοφληθεί το αμερικανικό χρέος από αύξηση των, της φορολογίας ή τέτοιων τακτικών μέτρων. Θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρετικά μέτρα. Θα διατηρήσετε, είναι πρόθεσή σας να συνεχίσετε το σύμφωνο ή θα συνεχιστεί η αναστολή του και θα οδηγήσει σε μια νέα χαλάρωση όπως ελέγχθη το 2005 ή μήπως θα το παραπέμψουμε ε, στις ρωμαϊκές καλένδες και θα το ξεχάσουμε μια και καλή το σύμφωνο σταθερότητας. Ποια είναι η πρόθεσή σας. Ποιο περιθώριο λιγμών έχετε δε ε, σε σχέση με την αναστολή του συμφώνου ε, τι, πώς πλήττει η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, την αξιοπιστία των δημοσίων οικονομικών. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Και το τρίτο σημείο, το πρόγραμμα ανάκτησης δημοσιονομικής ισορροπίας. Τι προτίθεστε να κάνετε από αυτό. Θα επιταχύνετε, θα αυξήσετε την πίεση ε, επί των κρατών μελών που έχουν έλλειμμα θα ζητηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτά. Η Λισαβόνα, επίσης πολύ σημαντικό ε, ε, στοιχείο. αφήνοντας να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα, ξέρετε Ισπανός είμαι, θα πρέπει να κάνω και μια παρομοίωση με Ταύρο δεν γίνεται αλλιώς. Από τα κέρατα λοιπόν να πιάσει τον τάβρο η Ισπανική Προεδρία μετά από εσά. Η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού δεν ε, αποδείχτηκε ο λίγων αποτελεσματική. Θα κάνετε κάτι από αυτού, ε, κυρώσεις για μη συμμόρφωση, ε, αλλαγή του συστήματος, έχετε κάποιες προθέσεις από αυτού. Και ένα πιο γενικό, για να μην πω φιλοσοφικό ερώτημα. Η νέα Λισαβόνα έχει δεκαετή ορίζοντα με τις προκλήσεις που έχουμε, ανταγωνιστικότητα, γύρανση του πληθυσμού, κλιματικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Μήπως θα πρέπει να έχουμε πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, όχι δεκαετή, αλλά πιο πολύ. Αυτά εκ μέρου μου. Ευχαριστώ τους δύο παρόντες ε, υπουργού. Η συνεργασία θα είναι όχι μόνο στενή, αλλά και απολύτως διασκεδαστική, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σεσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Πούλμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και από πλευρά μας θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε, να καλωσορίσουμε τους ε, εκπροσώπους της Προεδρία. Προεδρίας και εμείς ε, χαιρόμαστε και ελπίζουμε να είναι καλή η συνεργασία. Θα θέλαμε κυρίως σε τρία θέματα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας και να θέσουμε και κάποιες ε, απαιτήσει από πλευράς δηλαδή συνομοθέτη από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο έχει μεγάλο συμφέρον να βγει από την κρίση η οικονομική πολιτική μέσω της καλύτερης συνεργασίας. Αυτή η Επιτροπή ασχολείται με την νομοθεσία των χρηματοπιστωτικών αγορών και σήμερα συζητήσαμε και είπαμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι καλή η νομοθεσία. Ξέρουμε, να ξέρουμε τι κάνουμε. Να έχουμε better regulation, καλύτερη ε, ρύθμιση νομοθεσία, όχι απλά πιο γρήγορη νομοθεσία και θα θέλαμε παράλληλα να υπογραμμίσουμε το εξής. Πρέπει να υπάρχει καλή ρύθμιση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε, αν θέλετε, το θάρρος μας για να δημιουργήσουμε νέους κανόνες. Αυτό μας έμαθε η κρίση, ότι χρειαζόμαστε ένα νέο παιχνίδι, νέους κανόνες για το παιχνίδι. Να μην αφήσουμε να μας επηρεάσουν τα μεμονωμένα συμφέροντα, να μην μας εμποδίσουν τα μεμονωμένα συμφέροντα, να καταρτήσουμε μια σωστή νομοθεσία για την χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη. Να επιδείξουμε δυναμισμό δεύτερο στοιχείο το οποίο θέξατε και εσείς ο ίδιος, η κρίση στην εργασιακή αγορά, στην πραγματική οικονομία. Σε πολλές περιπτώσεις το να διδαχόμεθε από τις σκανδιναβικές οικονομίες σημαίνει το πώς μπορούμε να δημιουργούμε νέες αξίες για τον κάθε εργαζόμενο προκειμένου να έχουμε καλές συνθήκες για τις εργασιακές συνθήκες του αύριο και αυτό το εγγυάται και η Λισαβόνα 2. Ως Σουηδική Προεδρία είχατε δώσει κάποτε πολύ σωστά κίνητρα με τη διαδικασία της του Γκότεμπεργκ. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενθαρρύνουμε και πάλι να επιδείξετε την ίδια δημιουργικότητα, να αναλάβετε τέτοιο ηγετικό ρόλο και μαζί με την Ισπανική Προεδρία, την επερχόμενη Προεδρία, να φροντίσετε να δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά αυτή την ρύθμιση, να μην μείνουν όλα στα χαρτιά. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο. Μάθαμε από την κρίση πόσο δύσκολο και ατυχές είναι όταν η Ευρώπη διεθνώς δεν ομιλεί με μία φωνή. όσους σοσιαλιστές και δημοκράτες πρέπει να σας πω ότι σε κάθε ευκαιρία σας ενθαρρύνουμε είτε στους G20 ή σε διάφορες διασκέψεις για το κλίμα να αναφέρετε ότι η Ευρώπη όλο και πιο πολύ δρά από κοινού με μια κοινή στρατηγική προκειμένου οι άλλοι να καταφέρουν να συντονιστούν μαζί μας. Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουμε και αυτός είναι ο σκοπός που προσπαθούμε να πετύχουμε. Thank you. Ευχαριστώ. Σοφή και μετά θα δώσω το λόγο στην Προεδρία. Και απομένουν άλλες δέκα περίπου ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να τις μοιράσω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Σουηδική Προεδρία για την παρουσίασή της. Χάρηκα πολύ ακούγοντας την προσέγγισή σας γιατί το μήνυμα είναι αρκετά ανησυχητικό. Είπατε ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέσο έλλειμμα 7%. Δεν είδα κανέναν λιποθυμάει, αλλά είναι πολύ περίεργο αυτό το νούμερο και θυμηθείτε και το δημόσιο χρέος εδώ. Το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο 1,5 χρόνο θα μιλάμε αρκετά για την ε, ρύθμιση των αγορών. Τι θα γίνει όμως με τους δημόσιους φορείς. Γιατί δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι πολλές χώρες πριν την κρίση είχαν αδιαφορήσει για την το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τουλάχιστον μία χώρα μπορώ να σκεφτώ που το έκανα. Δεν πρέπει λοιπόν επιτέλους να βρούμε κάποιους τρόπους για την ε, συμμόρφωση και την επίβλεψη της συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ένα δεύτερο θέμα αφορά τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί τεράστια ποσά ως κρατικές ενισχύσεις και μας είχαν υποσχεθεί ότι όλα αυτά αφορούσαν την πράσινη ανοικοδόμηση, ότι επιτέλους μπαίνουμε στον 21ο αιώνα, ότι θα έχουμε καινοτομία. Ναι, αλλά τελικά αυτό που βλέπω είναι ότι τα περισσότερα χρήματα μπήκαν είτε στις τράπεζες είτε στις υπάρχουσες βιομηχανίες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τη Σουηδική Προεδρία αν ενδιαφέρεται να κάνει κάποιο είδου αξιολόγηση για να δει κατά πόσο αυτές οι κρατικές ενισχύσεις δόθηκαν όντω για μια πράσινη επανάσταση ή για μια επανάσταση καινοτομία. Επίσης, είπε και ο συνάδελφός σας ότι μάλλον θα καταλήξετε σε μια συμφωνία όσον αφορά τα μπόνους και τις, μισθού. Ε, τους Αυτό είναι πολύ καλά, αλλά θα γίνω κοινική εδώ. Μήπως όλα αυτά δεν είναι παρά βιτρίνα. Ναι, υπάρχουν διάφορα φαύλα, αν θέλετε, κίνητρα στον κόσμο. Πολλά από αυτά αφορούν και πολιτικούς. Το γνωρίζουμε αρκετοί από εμάς. Υπάρχουν λοιπόν πολλές προτάσεις αυτές τη στιγμή όσον αφορά τις ρυθμίσεις και δεν είναι όλες πιστικές. Έχει υποθεί και δημοσίως ότι αυτό μπορούσαμε να καταφέρουμε από πολιτικής άποψης. Και ο υπουργός της χώρας μου είπε ότι αντί να προσαρμόσουμε την κρατική ενίσχυση στο μέγεθος των τραπεζών θα προτιμούσε να προσαρμόσει το μέγεθος των τραπεζών στις ενισχύσεις και να τις ε, μειώσει σε μέγεθος προκειμένου να μην υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση. Ρωτώ λοιπόν, Πιστεύετε ότι αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το θάρρος να λάβουμε ριζοσπαστικά μέτρα θα μπορούμε να το κάνουμε στο μέλλον ή θα καταλήξουμε σε μια νέα κρίση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία σε αυτές τις πολύ σημαντικές αλλά και περίπλοκες ερωτήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά τα μέτρα στήριξης ε, και την αποτελεσματικότητά τους, ειδικά όσον αφορά την εποπτεία και παρακολούθηση. Να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ύδατα που δεν γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και να θυμηθούμε ότι η κατάσταση τον Φεβρουάριο ήταν πολύ προβληματική, αλλά τώρα βλέπουμε τουλάχιστον κάποια θετικά. Τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα είχαμε σταθεροποίηση, τουλάχιστον όσον αφορά την χρηματοδότηση από τις τράπεζες που πλέον βρίσκεται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά πριν την κρίση. Βεβαίως για την τελική αξιολόγηση θα πρέπει να περιμένουμε ένα-δύο χρόνια τουλάχιστον. Πάντως τόσο η Κεντρική Τράπεζα όσο και οι κυβερνήσεις προχώρησαν άμεσα σε μία πολιτική που έδωσε λύσεις. Τώρα, όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας, θεωρώ ότι κινούμαστε εντός του Συμφώνου Σταθερότητας, γιατί υπάρχει κάποιος βαθμός ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Και είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση. Βεβαίως υπάρχουν πολλές πολύ προβληματική αριθμή σε αρκετές χώρες. Αύξηση της ανεργίας, μείωση της ανάπτυξης ε, και της παραγωγής. Άρα βρισκόμαστε σε μια τυπική περίπτωση όπου πρέπει η φορολογική πολιτική να αναλάβει σταθεροποιητικό ρόλο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδαμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Τώρα όμως πρέπει να το δούμε και ευρέως το θέμα, να δούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στην αγορά απασχόλησης και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι παραγωγικές μας δυνατότητες μπορεί να πληγούν στο μέλλον. Και επίσης πολλές βιομηχανίες αυτοκινητοβιομηχανίες και τα λοιπά, είναι άγνωστο αν θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες παραγωγής στο μέλλον. Αυτά είναι θέματα δομικά τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Υπάρχει η φορολογική πολιτική που μπορεί να μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα στο θέμα της ανεργίας. Γνωρίζουμε τι είχε γίνει τη δεκαετία του 70 με τα σοκ της ανεργίας και την άνοδο σε τρομερά επίπεδα της ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα να έχουμε υπόψη μας και μια μελλοντική αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και αποδοτική. Για να απαντήσω στον κύριο Πούλμαν τώρα. Ναι, χρειαζόμαστε καλή νομοθεσία στην Ευρώπη. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος όταν αντιμετωπίζουμε κρίσεις ότι προχωρούμε υπερβολικά γρήγορα. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι προχωρούμε υπερβολικά αργά, καθυστερημένα. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα να πούμε σε μία χώρα ότι αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη κρίση μετά την το κράχ του 29 και να τους πούμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βεβαίως πρέπει να βρούμε νομοθεσίες οι οποίες θα είναι πιο ευρείες και πιο λογικές και επιφυλεκτικές. Πρέπει να διδαχθούμε από την κρίση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε πιο ευρεία, πιο αυστηρή, πιο συνετή νομοθεσία. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Ο κύριος Μπούλμαν μας μίλησε για την κοινή φωνή της Ευρώπης. Όντως προσπαθούμε να το κάνουμε στα πλαίσια του G20 και προσπαθούμε να το κάνουμε και για τις λύσεις που θα προτείνουμε στην Κομπεχάγη. Όμως σκεφτείτε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια διαδικασία όπου θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε απλά μία φωνή. Θέλουμε μία φωνή η οποία θα είναι νομιμοποιημένη και θα προκύπτει από μία σωστή και εμπεριεκτική διαδικασία. Η κυρία Ιντερφέλτ, ο κύριος Κλίνς είπε κατά λάθος ο Υπουργός, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό και η Αμερική αντιμετωπίζει τα ίδια θέματα. Και βεβαίως να πω ότι η πρόβλεψη της Κομισιόν είναι για 7 με 8% έλλειμμα μετά την κρίση. Γιατί θεωρούμε ότι θα έχουμε κατά μέσο όρο 25% αύξηση του δημόσιου χρέους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Βεβαίω, τα προβλήματα του χρέου, τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού και τη ανεργία υπήρχαν και πριν την κρίση, αλλά τώρα εντείνονται. Άρα μας αναμένει δύσκολο έργο, ειδικά σε θέματα της διαδικασίας της Λισαβόνα. Και ναι, χρειαζόμαστε δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, όπως για παράδειγμα την αύξηση της ανεργίας και την αρνητική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας στην φορολογική πολιτική, κάτι που θα έχει και βραχυπρόθεσμες θετικές συνέπειες. Βεβαίω, γνωρίζω ότι οι διαδικασίε ε, στην ε, Ολλανδία είναι αυστηρέ και καλές και το ίδιο ισχύει και για τη Σουηδία. Πρέπει να ισχύσει σε όλες τι χώρε. Ναι, δεν υπάρχει το κοινό πλαίσιο του Συμφωνού Σταθερότητας, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί με αυστηρό τρόπο. Και αυτό έχει να κάνει με τους εθνικού προπολογισμού βεβαίω. Βεβαίως θα ασχοληθούμε με τις όποιες υπερβολές στο θέμα της, του Συμφώνου Σταθερότητας. Θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή. Υπάρχει και η συνάντηση στο Γκέτεμπορκ φέτος στο φθινόπωρο. Δεν πρόκειται λοιπόν να το γνωρίσουμε. Τώρα όσον αφορά την πράσινη ανάκαμψη η δική μου κυβέρνηση είναι πολύ επιφυλακτική. Δεν θεωρούμε ότι είναι αποδοτικές ε, οι ενισχύσεις συγκεκριμένων βιομηχανιών. Όμως, από την άλλη πλευρά, θυμηθείτε ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το πώς θα είχαμε μία συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και ένα ισότιμο πεδίο για όλους. Θέλαμε να έχουμε γρήγορη και συστημική αντίδραση. Ναι, θα μπορούσε να έχει έρθει η Deutsche Bank και να μας πει ότι εμείς θα χρηματοδοτήσουμε τη Volvo. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ευελιξία στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων Τώρα, όσον αφορά τα πόνους, δεν νομίζω ότι είναι απλά θέμα βιτρίνας. Ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα αυτό, ότι αν επιβραβεύεται όσους λαμβάνουν υψηλούς κινδύνους, τότε θα το κάνουν ακόμη περισσότερο. Και υπήρχε μία ασυμμετρία εδώ, γιατί υπήρχαν μεγάλες επιβραβεύσεις σε πολλές περιπτώσεις και όχι κάτι αντίστοιχο στις περιπτώσεις που δεν απέδιδαν αυτή η κινδύνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία πιο ισορροπημένη θεώρηση των θέματος των πόνους. Επαναλαμβάνω, σε όλους τους νέους ε, μας ε, κανονισμούς και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να είμαστε ευρείς, αυστηροί και συνετοί. Βεβαίως δεν πρόκειται να αποφύγουμε μια επόμενη κρίση. Έχουν υπάρξει και πολλές κρίσεις στο παρελθόν, .com και τα λοιπά. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε καλύτερα. Thank you for all. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τις επικοδομητικές σας ε, παρατηρήσεις και για την υποστηρίξή σας και την ενθάρρυνσή σας να συνεχίσουμε αυτά που έχουμε ξεκινήσει. Απάντησε ο συνάδελφος ήδη σε πολλές ερωτήσει. Θα ήθελα να πω ότι η βασική εισρωή ρευστότητας που έγινε από διάφορες τράπεζες έγινε με το σωστό τρόπο και επίσης ήταν πολύ επικερδής για τις τράπεζες αυτές. Έβγαλαν μεγάλο κέρδος. Νομίζω ότι ήταν λοιπόν μια εύστοχη διαδικασία χωρίς την οποία θα είχαμε πραγματικά μια κατάρρευση, μια πλήρη κατάρρευση. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πραγματικά κάτι ωφέλιμο. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι από, το, από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στις διάφορες χώρες και κυρίως και στη δική μας χώρας, χώρα αλλά και στις δικές σας χώρες. The core here. I think we need crystal clear... Η βιτρίνα. Για τη βιτρίνα, το θέμα της βιτρίνας. Τι χρειαζόμαστε. Καθαρούς και ξεκάθαρους κανόνες. Με εποπτεία και με κυρώσεις για τις τράπεζες οι οποίες θα παραβιάσουν τους κανόνες αυτούς. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το στόχο μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο G20. Ευχαριστώ. Ναι, λυπάμαι που σας διέκοψα, λέει η Πρόεδρος, αλλά δεν μπορούσα να δω πώς θα τους χωρέσω όλους. Καλή ιδέα θα ήταν να ακούσουμε λοιπόν έξι ομιλητές, προτού απαντήσετε. Και μετά να απαντήσει η Προεδρία. Okay. Σας ευχαριστώ και για να είμαστε σύντομοι. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένη για την οδηγία για τους διαχειριστές των ελλακτικών επενδυτικών μέσων. Αυτό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Μπορέσατε να συλλέξετε δεδομένα για το πού μπορεί να υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι ή αν θέλετε ενδεχόμενοι συστημικοί κίνδυνοι. Μπορεί να μην θέλετε να μας το πείτε, αλλά από ό,τι κατάλαβα η ομάδα σας προτιμάζει κάποιες βασικές ε, τροπολογίες ε, του κειμένου το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Αν αυτό αληθεύει θα ήθελα να δω τις ε, προτάσεις αυτές σύντομα. Φιλίπ. Okay, uh, Ναι, να κάνω λίγα σχόλια. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Προεδρία για την πρώτη πτυχή που ανέφερε, την εποπτεία. Θέλετε να υπάρχει εκτεταμένη εποπτεία, η οποία θα είναι και εφαρμόσιμη και θα εφαρμόζονται μάλιστα με τι αντίστοιχε κυρώσει. Έχετε δίκιο. Και συμφωνώ επίσης για το ότι κάθε παράγοντας στον κλάδο αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται, να τηρεί μάλλον τους κανόνες αυτούς. Τώρα, οι ανησυχίες ε, που μας διακατέχουν εμά ω Ευρωπαίους Πρασίνους. Επί του παρόντος, η πρόταση που έχουμε μπροστά μας προτείνει ουσιαστικά μια συντονισμένη δράση προς την ε, ρύθμιση και όχι ένα ενοποιημένο εποπτικό σώμα. Και αυτό μας απασχολεί. Είναι σαν να καταπολεμούμε τη μαφία με την τοπική αστυνομία. Συντονισμός, με συντονισμό με το τηλέφωνο, με τα email. Μιλάμε δηλαδή για συντονισμό και όχι για ενοποίηση. και εκεί υπάρχει μια έλλειψη σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Όντω, δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε μια φούσκα με μια άλλη, ένα κενό με ένα άλλο κενό. Να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι όντω ε, αναπτύσσεται και διωγγώνεται το δημόσιο χρέος και αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου και μιλάμε για ένα είδος χρέους αλλά υπάρχει και το χρέος το περιβαλλοντικό το χρέος ε, της εξάντλησης των πόρων και προφανώς το δημοσιονομικό χρέος δεν πρόκειται φυσικά να ωφελήσει τις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε όμως να κοιτάμε μόνο το ένα μέρος της εξίσωσης και δεν είναι ευχάριστη αυτή η πραγματικότητα γιατί δεν υπάρχει οποιαδήποτε εύκολη λύση στο δίλημα αυτό αλλά δεν υπάρχουν, θα πρέπει να βρούμε μια λύση για την εργασιακή αγορά μου προξενήσατε κάποια έκπληξη γιατί ο συνάδελφός σας ο ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας είπατε ότι η πρώτη γραμμή άμυνας θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κρίσης. Συμφωνώ. Δεύτερη γραμμή άμυνας είναι οι εργασιακές ε, συνθήκες, η εκπαίδευση. Και θα περίμενα να πείτε ότι υπάρχει και μία ενδιάμεση γραμμή η πράσινη μεταρρύθμιση, η δυνατότητα για την οικονομική δραστηριότητα που υπάρχει στην πράσινη ανάπτυξη. Και το ακούσαμε αυτό στην Επιτροπή Βιομηχανίας και θα περίμενα από την Σουηδική Προεδρία να είναι λίγο πιο συνεκτική. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες και σε ό,τι αφορά τις ε, εργασιακές πολιτικές της ενεργούς αγοράς. Να σας συστήσω προσοχή, να μην αποστείλουμε μηνύματα τα οποία θα κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι θα περιορίσουμε το επίπεδο της ασφάλειας. Γιατί αυτό τι θα σημαίνει, ότι ακόμα και όσοι έχουν θέσεις εργασίας θα είναι πιο προσεκτικοί με τα έξοδά τους και τις δαπάνες τους και αυτό φυσικά θα αποτελέσει ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα για τη μείωση της ζήτησης. Αν το κάνετε λοιπόν από αλτροιστικούς σκοπούς, να προσέξετε, γιατί υπάρχει και η πρακτική πλευρά του θέματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο το φορολογικό, σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς παραδείσους, δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις τις οποίες αποσκοπείτε να εφαρμόσετε. Και τέλος, για το να μιλάμε με μια ενιαία φωνή και συμφωνώ με τον συνάδελφο Μπούλμαν. Είσαστε αρκετά βέβαιοι ότι στην, ε, στο G20 οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλήσουν με μία φωνή. Είστε βέβαιος όμως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το χρέος και τις δημόσιες δαπάνες, γιατί δεν ακούω ακριβώς τα ίδια λόγια από πλευράς Γερμανίας και Γαλλίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάγεν. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τη Συνδική Προεδρία, η οποία πραγματικά δεν έχει εύκολο έργο. Νέο Κοινοβούλιο, νέα Επιτροπή Οσονούπο και βρισκόμαστε εν το μέσο της αντιμετώπισης της ε, κρίσης και εδώ και χρόνια συζητούμε για την απαραίτητη ρύθμιση και σήμερα το πρωί μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός πόσο σε δύσκολες και συγκρατημένες ε, ήταν ε, οι δηλώσεις ε, των Αμερικανών σε ό,τι αφορά δηλαδή τη ρύθμιση και τον καπιταλισμό. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε πιο πολύ ρύθμιση και το τονίζω αυτό γιατί αυτό αποτελεί ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σουηδική Προεδρία θα πρέπει να προσπαθήσει να διατυπώσει ομοιόμορφες ε, απόψεις εκ μέρους των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά θεωρώ ότι αυτό έχει και τα όρια του. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, στα πλαίσια των διαβολεύσεων για το πρόγραμμα της Μελλοντικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα αυτά θα γίνουν υπό Σουηδική Προεδρία, σας παρακαλώ λοιπόν να μεταβιβάσετε τις ε, απαιτήσεις μας αυτές προς τον νέο Επίτροπο. Θέλουμε σαφή ρύθμιση και το λέω αυτό εξ ονόμαστος της ομάδας μας παρά από τις διάφορες ε, φωνές που ακούγονται από τους φιλελεύθερους, από τους Ιρλανδούς και τους Βρετανούς. Ε, πρόκειται να ελέγξουμε πολύ αυστηρά το μελλοντικό Επίτροπο για να μην ε, ακολουθήσει την πολιτική του Μακρύβη. Και παρακαλώ την Σουηδική Προεδρία Είπατε μία πρόταση που μου έκανε το σκεφτώ αυτό. Είπατε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να δράσουμε υπερβολικά γρήγορα. Αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικά τόσο ελάχιστος. Ο αντίθετος κίνδυνος επικρατεί. Να δράσουμε υπερβολικά καθυστερημένα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο που θα ανοίξουν οι ΙΠΑ. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό τρόπο αντιμετώπισης και ρύθμισης. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτή η ελευθερία που συνεπάγεται το σύστημα αυτό ε, ακολουθήθηκε χωρίς να υπάρχει συνέστηση και της υποχρέωσης, της ευθύνης που τη συνοδεύει την ελευθερία αυτή. Σας παρακαλούμε λοιπόν, γιατί μάλλον να συμμετάσχετε στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση τη χρηματοπιστωτική. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Κοινοβούλιο να υπονομευτεί όπως τα τελευταία πέντε χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν σας απευθύνω την εξή έκκληση. Να εξετάσετε με πάσα σοβαρότητα όπως απευθύνθηκε και έκκληση και στον ε, Σουηδό Πρωθυπουργό. πότε και αν η Σουηδία θα γίνει μέλος της Ευρωζώνης. Γιατί δεν έχετε πολιτική διέξοδο, έχετε πολιτικές ε, αποφάσεις τις οποίες δεν επιθυμείτε ίσως, αλλά θα πρέπει να καταστείτε επιτέλους μέλος της Ευρωζώνης. Και καλό λοιπόν την Σουηδική Προεδρία να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Thank you. Ευχαριστώ, Καθρίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. δεν μιλάμε, δεν είναι σωστό να μιλάμε για βρετανικό, ιρλανδικό ή αμερικανικό πρόβλημα. Όλοι μαζί ε, στο ίδιο καλάθι βρισκόμαστε και επιτυχίες ε, όλοι θα πιστοθούμε αν επιτύχουμε, αποτυχίες όλοι θα χρεωθούμε αν αποτύχουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτά που είπε για την ε, στρατηγική της Λισαβόνας αυτό που λέγαμε για την ε, ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου που θα βασίσεται στη γνώση και που θα έχουμε επιτύχει μέχρι το 2010 πόρο απέχουμε. Ο στόχος είναι πολύ σωστός, αλλά κάπου κάναμε λάθος. Κοιτάξτε τι γίνεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι Yahoo, τι Amazon, εμείς τι κάναμε εδώ. Πώς καινοτομήσαμε. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Χαίρομαι λοιπόν που θέσατε το θέμα αυτό και για τις κλιματικές αλλαγές. Εγώ κατά την προεκλογική περίοδο μίλαγα πάντα για πράσινη απασχόληση, για πράσινη ανάπτυξη και όλα τα πολιτικά κόμματα σε όλο το φάσμα αλλά έχουμε μείνει σε λόγια, πολύ φοβούμε. Σε έργα δεν έχουμε ακόμα περάσει. Και για την έκθεση που αναφέρατε για την ε, Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ε, του Λονδίνου, πολύ θα ήθελα να τη διαβάσω γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Τώρα, για την πρόταση για την εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία και αυτό που είπε ο συναδελφός σας για κατάλληλη νομοθεσία για τους φορείς εκείνους του συστήματος ε, που ε, αποτελούν κίνδυνο. Μιλήσατε για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα, για τις ε, πληροφορίες που θα πρέπει να ελέγχονται κτλ. Το βασικό ζήτημα πιστεύω είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία προσέγγιση unisex. Άλλοι μιλάνε για τα hedge funds, άλλοι μιλάνε για τα private equities, άλλοι για τις ε, επενδυτικές, ε, ε, για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που θα πληγούν από αυτό το νέο σύστημα και που δεν ευθύνονται σε τίποτα για την αναφύγηση της κρίσης. Λοιπόν, όχι unisex. Κάθε πρόβλημα έχει τη δικιά του λύση παρότι το πλαίσιο είναι κοινό. Βέβαια δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Οι στόχοι που αναφέρατε δεν ξέρω αν θα ε, επιτευχθούν. Αλλά κάλιο ένα και στο χέρι λέμε εμείς ε, παρά πέντε και καρτέρι. Και είναι σίγουρο ότι η Ιρλανδία θα είναι στις συνθήκες της Λισαβόνας πριν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ καλό αυτό το τελευταίο που είπατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, είπε και ο κύριος Λάγκερ, χρειαζόμαστε ρυθμίσεις όντως, αλλά όχι τόσες πολλές. Δηλαδή να μην ε, επιβάλλουμε ρυθμιστικές διατάξεις που είναι αντιπαραγωγικές. Αυτό ήταν αυτό που ήθελα να πω και τώρα περνάω στη μητρική μου μια που απευθύνομαι και στην Σουηδική Προεδρία. Δύο υπουργούς κέντρο δεξιάς συμμαχίας, δεξιού συνασπισμού έχουμε εδώ. Αυτό με ε, ευχαριστεί ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κανένα σοσιαλδημοκρατικό στοιχείο στην αντιπροσωπεία αυτή. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θέτω ένα ερώτημα ως Σουηδός πολίτης. Η Σουηδική οικονομία θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καλύτερο ήταν να είναι εκτός του ευρώ όταν επλήγημεν από την κρίση. Στο Παρέσι αποφασίστηκαν μια σειρά σημαντικών θεμάτων και τότε πάλι δεν θέλατε να θίξετε το θέμα της Ευρωζώνης τώρα με τη στερνή γνώση. Τι πιστεύετε, καλύτερα εντός ή καλύτερα εκτός. Και πότε θεωρείτε, αν αποφασίσετε ότι θέλετε να είστε εντός, ότι θα τα καταφέρετε. Τώρα, για τον Υπουργό Ντελ. Παρακολουθώ τις δηλώσεις σας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. η αρμοδιότητά σας είναι πλέον έχει μεγαλύτερη σημασία διότι προεδρεύεται των Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σουηδία όμως είναι μια μικρή ανοιχτή χώρα προσανατολισμένη προς τις εξαγωγές. Υπάρχουν άλλες χώρες με ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά. Πώς θα μπορέσετε να τα συμφιλιώσετε όλα αυτά. Πώς θα έχετε ισορροπημένη παρουσίαση των συμφερόντων της Ένωσης. Είπε ο κύριος Σοντέλ ότι υπάρχει αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση, αλλά ελπίζω ο κύριος Σοντέλ θα αποφύγει την παγίδα της ρητορία που χαρακτηρίζει τις δηλώσεις ηθινόντων από χώρε όπως η Γερμανία ή η Γαλλία και θα έχει πρακτική μέρημνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλέντερ, ναι, μία ερώτηση έχω να απευθύνω προς τον κύριο Μπόρκ. Είπατε πριν από λίγο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει με μία φωνή. Ναι, να επαναλάβω. Είπατε ότι η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με μία φωνή. Και στην σύνοδο του G20. Στις αρχές της εβδομάδας η κυρία Μέρκελ ο καγκελάριο και ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή ανέφεραν ότι θα πρέπει να ε, περιοριστούν οι αμοιβέ των ε, τραπεζικών στελεχών ως μέτρο ρύθμισης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας θέση. Συμφωνείτε, γιατί είναι σημαντικό φυσικά αυτό για να μιλήσει η Ευρώπη με μία φωνή. Δεύτερη πτυχή τώρα. Μιλώ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Συμφωνούμε απόλυτα με την εκτίμηση ότι η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών θα πρέπει να βελτιωθεί. Ωστόσο, δεν συμφωνούμε με την εκτίμηση ότι η εποπτεία δεν αποτελεί τμήμα του προβλήματος. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα είναι πιο βαθιά. Δεν είναι μόνο θέμα εποπτείας, πρόκειται για θέμα κανονισμού ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την ίδια την ουσία της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών και να την τροποποιήσουμε. Και αυτό σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη, να μην περιοριστείτε δηλαδή μόνο στο επίπεδο της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και μια τρίτη παρατήρηση. Την Το προηγούμενο Σαββατοκυριακό άλλαξε η κυβέρνηση στην Ιαπωνία. Είχαμε εκλογέ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μελλοντική, η επερχόμενη Ιαπωνική κυβέρνηση ανέφερε ότι δεν θα επικεντρωθεί πλέον στις εξαγωγές θα επικεντρωθεί στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για μια αλλαγή των πολιτικών και οικονομικών ε, ε, προοπτικών. Ποια είναι η δική σας στάση και ιδιαίτερα εν ώψη και της στρατηγικής Λισαβόνας, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στις εξαγωγές. Uh, Ολοκληρώσαμε με αυτήν την δέσμη ερωτημάτων. Έχουμε ακόμα έξι ομιλητές και 25 λεπτά της ώρας στη διάθεσή μας. Θα είμαι σύντομος λοιπόν στις απαντήσεις μου και ο κύριος Οντέλ θα με συμπληρώσει. Για τον Φίλιπ Λάμπερτς, για τα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο χρέος και πώς ε, σχετίζεται με το περιβαλλοντικό χρέος. Δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Δεν βλέπω γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε και τους δύο στόχους και η Δανία και η Σουηδία μπόρεσαν να έχουν ε, ε, φιλικά ε, επί του περιβάλλοντος μέτρα, μείωση του δεξιδίου του άνδρα των εκπομπών κτλ. χωρίς να έχουν οικονομικές ζημίες στα δημόσια οικονομικά τους. Ορισμένες από αυτές τις λύσεις που προκρίναμε βοήθησαν και για την επίλυση του δημοσιονομικού χρέους ελλείμματος, του δημόσιου χρέους τέλο πάντων, αλλά και του περιβαλλοντικού χρέους. Και νομίζω ότι βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά μπορούν και, τα, και οι δύο στόχοι να επιτευχθούν. Και η φορολόγηση της ενέργειας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε όταν προκύψει σχετική πρόταση της Κομισιόν. Τώρα, ει ό,τι φορά τι γραμμέ αμήνη που ανέφερε ο κ. Ναι, όντω, η πρώτη γραμμή είναι η δημοσιονομική άμυνα. Η δεύτερη γραμμή είναι η ζήτηση. Να προλάβουμε τη μείωση της ζήτησης. Παράλληλα, αυξάνοντας την απασχόληση και μειώνοντας την ανεργία. Και η τρίτη γραμμή άμυνας είναι διαρθρωτική άμυνα, προληπτική αν θέλετε. Να μην επιτρέψουμε στην ανεργία να αυξηθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ενεργούς πολιτικές. Να δώσουμε κίνητρα. Η εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο, η παιδεία, αλλά και σωστές αμοιβέ. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι υπάρχουν διαταραχές στην αγορά απασχόλησης και αυτό οδήγησε σε πολλά προβλήματα ανεργίας γιατί υπάρχει πρόβλημα αμοιβών. Φοροδιαφυγή. και ισοτιμία μεταξύ των, ε, δημοσιονομικών αγορών. Ναι, είναι στόχος μας. Θέλουμε να εργαστούμε από αυτού. Και γι' αυτό ετοιμάζουμε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση. Και ενώψη του Λονδίνου και ενώψη του Πίτσμπεργκ. Ο κύριος Λάγκεν ανέφερε τις προσδοκίες του για το G20. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος στην άτυπη συνάντηση που είχαμε σήμερα, πιστεύω ότι πραγματικά μπορέσαμε να καταλήξουμε στις αδρές, αν μη τι άλλο, γραμμές μιας κοινή θέσης για τις αμοιβέ, τις αποζημιώσεις και τα μπόνους. και για το, κλιματι... για το θέμα των κλιματικών αλλαγών εν της Κοπενχάγης. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θέτουμε το ζήτημα κατά αντιμολία από τη μία δηλαδή ελευθερία, από την άλλη ευθύνη. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ευθύνη. Η ελευθερία δεν είναι αντίθετη, δεν είναι αντώνυμο της ευθύνης και τα δύο θα πρέπει να ενισχυθούν. Ο κύριος Στήλερ για την ε, στρατηγική της Λισαβόνας. Η κυρία Στήλερ για την ακριβία. Όντως, πόρο έχουμε από το στόχο. αλλά έχουμε και περισσότερα προβλήματα από τους Αμερικανούς ας πούμε διαρθρωτικής φύσεως πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της αγοράς απασχόλησης πρέπει να ενισχύσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις μεγαλύτερο επιχειρηματικό πνεύμα μεγαλύτερες επενδύσεις στην παιδεία, στην έρευνα στην καινοτομία μια πιο μακροπρόθεσμη και διαρθρωτική θεώρηση των πραγμάτων θα καταλήξουμε σε κάποιο είδου πολιτική συμφωνία το Δεκέμβριο και θα δώσουμε τη σκητάλη στην Ισπανική Προεδρία να προχωρήσει περισσότερο τα πράγματα. Συστημική κίνδυνη. Ούτε τα hedge funds, ούτε τα private equities ήταν το πρόβλημα. Το κεφάλαια ήταν το πρόβλημα, τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια και στον πυρήνα της, στην καρδιά της ρωσικής κρίσης το 98 κεφάλαια δεν υπήρχαν. Και οι Αμερικανοί με τους ε, Lehman Brothers κεφάλαιο δεν είχαν. Ναι λοιπόν ότι ένα κομμάτι του προβλήματος είναι ε, ότι δεν υπήρχε αρκετή ρύθμιση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια πιο αυστηρή ρύθμιση είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική. Για τα σχόλια σας για την Σουηδία και την Ευρωζώνη. Ο Ντέγκ Τσαοπίνγκ για την Γαλλική Επανάσταση είχε πει «Οψόμεθα, είναι ακόμα νωρίς να σχολιάσουμε». Δεν θα πω αυτό κι εγώ. Είχαμε δημοψήφισμα Όλοι οι ηγεσίε των πολιτικών κομμάτων είναι υπέρ και συμφωνήσαμε ότι θα περάσουν τουλάχιστον 10 χρόνια μέχρι να ξανανοίξει το ζήτημα. Είναι πιο δημοφιλές το ευρώ από ό,τι ήταν παλιά που θεωρείται πυλώνας της σταθερότητας στα χρόνια αυτά της κρίσης. Η κοινή γνώμη είναι όμως επιφυλακτική. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και την αίσθηση της κοινή γνώμης. Ναι, αλλά υπάρχουν και νομοθετικά προβληματάκια, ξέρετε, που θα πρέπει να επιλύσουμε και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε από την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία ε, για να μπούμε στο ευρώ. Όσες φορές και αν ψηφίσω εγώ, ναι, δεν αρκεί. Για την πρωτοβουλία Μέρκελ, θετικότατη. Η συνάντηση που είχαμε σήμερα στο Συμβούλιο μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις της Καγκελαρίου δίνουν νέα όθηση στη συμφωνία αυτή και νέα ορμή στην θέση μας εν και του Λονδίνου και του Πίτσμπεργκ. Σε πλαίσια, στα πλαίσια της Τρόικα και με την Γαλλία και με την Ισπανία αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά και είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το αναφέρω. Τώρα για τις αγορές έχω διαφορετική άποψη από εσάς, διαφωνώ με αυτό που είπατε και το τελευταίο είναι ότι η χώρα μου είναι όντως η, από τις πιο προσανατολισμένες στις εξαγωγές. Ε, είμαστε αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την παραγωγή μας, βελτιώνουμε την ταχύτητα εξάπλωσης των νέων τεχνολογιών πιο εύκολα. Ε, το μοντέλο μας ε, πιστεύω ότι μας δίνει μια, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και δεν το αμφισβητώ επουδενή. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η κυρία ρώτησε αν ήδη συλλέγουμε δεδομένα για, την, ε, για τον εντοπισμό των συστημικών κινδύνων. Ναι, γίνεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις ε, Εθνικές ε, αρχές της FCA. Βεβαίως η τελευταία φορά είχε γίνει το 2001 για την Σουηδία, τότε που ήταν και η αρχή της διαδικασίας Λαμφαλουσί. Όμως τότε δημιουργήθηκε ένα ισότιμο πεδίο για όλη την Ευρώπη και αυτό ήταν ιδιαίτερα καλό. Όμως το κακό είναι ότι παραμείναμε σε εθνικό επίπεδο. Τώρα όμως η διαδικασία λαμφαλουσί είχε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε διαβούλευση, θα μάθουμε νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη Σεπτεμβρίου με πέντε νομοθετικές προτάσεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα επί Σουηδικής Προεδρίας. Αυτό είναι ο στόχος μας. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα, ο κύριος Λάμπερτ ζήτησε λιγότερο συντονισμό και περισσότερες πρωτοβουλίες. Πρέπει να δούμε τι είναι πολιτικός δυνατόν. Τώρα έχουμε για παράδειγμα τις τρεις αρχές σε μικροεπίπεδο. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, βρίσκει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ολοκλήρωσης και συντονισμού. Ναι, οι τράπεζες πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει όμως να υπάρξει συνεργασία και συντονισμός. Επαναλαμβάνω και αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σας. Πάντως να πω ότι εγώ θα ψηφίσω ναι στο επόμενο δημοψήφισμα για το ευρώ. Θα απαντήσω στα σουηδικά στον κύριο Σμιτ. Α, βλέπω και άλλο παλιό φίλο, τον κύριο Χοικμάρκ, στην αίθουσα. Πολιτικά όλοι μάλλον συμφωνούμε ότι θα ήταν καλύτερα να ήμασταν στο ευρώ. Όμως η Σουηδία εξαρτάται από τις εξαγωγές της. Αυτή τη στιγμή στην κρίση εμείς ευνοηθήκαμε στις εξαγωγές μας. Μας ήταν πιο εύκολο να κάνουμε εξαγωγές με ασθενέστερο νόμισμα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει εκ των υστέρων να εξετάσουμε και να καταλήξουμε στο αν ήταν θετική ή αρνητική η απουσία μας από το ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όσον αφορά την οδηγία για τις εναλλακτικές επενδύσεις περιλαμβάνει μια πολύ ανομοιογενή ομάδα επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά όλες τις νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες και να δούμε πού επιτυγχάνουν όντως το στόχο τους οι προτάσεις, πού θα έχουν θετικές συνέπειες να πω ότι χαίρομαι γιατί ήδη έχουμε δει πρόοδο τόσο στην ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο όσο και στις συζητήσεις μας με τη βιομηχανία που πλέον είναι πολύ πιο επικοδομητική. Πιστεύω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο, μια καλύτερη νομοθεσία που δεν θα δημιουργεί επιπλέον άχθος για τη βιομηχανία, αλλά παρόλα αυτά θα ρυθμίζει καλύτερα αυτή την αγορά. Γιατί δεν μπορούμε να την αφήσουμε χωρίς ρύθμιση αυτή την αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Οι τελευταίοι έξω μιλητές. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί δεν θα προλάβετε να ακούσετε τις απαντήσεις. Γκέρι, εκτός μικροφώνου. Με συγχωρείτε. Θα μιλήσω γκρικά. όπου σύμφωνα με το νέο γλωσσικό νόμο της Σλοβακίας, αν είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα στη χώρα της Σλοβακίας, θα αντιμετώπιζα σοβαρές επιπτώσεις. Όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας, οι Υπουργοί ανέφεραν ότι χρειάζεται διαφάνεια στις ρυθμίσεις. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλλά επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Δύο πράγματα λοιπόν δεν μπορούμε να αγνοούμε. Καταρχάς, οι πολίτες μας μπορεί να αναρωτηθούν και με το δίκιο τους αν είναι αξιόπιστοι όταν εγκρίνει κανόνες που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. ακούνε ότι η διαδικασία υπερβολικού ελίματος θα είναι αναπόφευκτη για όλες είναι τα κράτη-μέλη. Ρωτάω λοιπόν τη Σουηδική Προεδρία. Έχετε κάποια πρόταση επ' αυτού προκειμένου να αποφύγουμε την είσοδο σε ένα φαύλο κύκλο γιατί από τη μία χρειαζόμαστε ανάπτυξη και από την άλλη με αυτά τα υπερβολικά ελλείμματα θα είναι σχεδόν αδύνατο. Έχετε κάποια λύση να προτείνετε λοιπόν. Ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε την επιτρεπόμενη διαφορά στο δημόσιο έλλειμμα. Και ίσως θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε τον το όριο για τον πληθωρισμό με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της και όχι τη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι η συνεργασία σας μαζί μας θα είναι τόσο καλή όσο και στο παρελθόν με άλλες προεδρίες. Έχω διάφορες ερωτήσεις, αλλά έχω να σας προσφέρω και τη βοήθειά μου. Συμμετέχοντας στην διαδικασία G20, κάνετε ένα σημαντικό βήμα προς το εμπρός. μας λέτε ότι δεν εντοπίζετε κάτι που αντιτίθεται στα συμφέροντα της Ένωσης. Σας ρωτώ όμως τι μπορεί να κάνει για να σας βοηθήσει το Κοινοβούλιο προκειμένου όντως να μιλήσετε με μία φωνή στην G20. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Χαίρομαι που σας βλέπω και νομίζω ότι είναι καλό που έχουμε Σουηδική Προεδρία σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική θητεία και καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα εκτός κρίσης. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη κρίση. Γιατί πάντα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε προβλήματα, το δύσκολο είναι να βγούμε από τους πελάδες θα συζητήσουμε αρκετά το θέμα της καλύτερης ρύθμισης των αγορών. Πρέπει όμως να δούμε και το θέμα της καλύτερης ρύθμισης των μακροοικονομικών μεγεθών. Στο παρελθόν αλλάξαμε το σύμφωνο σταθερότητας μειώνοντας την ελαστικότητα, όμως ίσως θα έπρεπε να την αυξήσουμε τουλάχιστον για προβληματικές περιόδους. Ε, κάτι που ξεχνάμε είναι ότι ορισμένες χώρες είχαν μεγάλα ελλείμματα και πριν την κρίση. Κάτι που σημαίνει ότι ήταν λιγότερο προετοιμασμένες για την κρίση. Προκύπτει λοιπόν μια συζήτηση για το τι θα έπρεπε να ισχύει όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τα ελλείμματα σε καλούς καιρούς. Και πρέπει να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση γιατί διαφορετικά ποτέ δεν πρόκειται να την συνεχίσουμε. Όχι σίγουρα όταν θα βρισκόμαστε εντός της κρίσης. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο ερώτημα. Η ανεργία έφτασε στο 9,5% ε, στην Ευρωζώνη είναι όντως ε, ο δείκτης αυτός έχει κάποια ε, ε, σχετική αξία. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να λέμε ότι βαδίζουμε στον καλό δρόμο όσο συνεχίζεται να αυξάνεται η, η ανεργία. Δεν θεωρεί η Σουηδική Προεδρία ότι θα πρέπει να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα από τη μέχρι τώρα ένα πραγματικό πρόγραμμα ανάκαμψης ε, ζωογόνησης των επενδύσεων, των ε, διαρθρωτικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης. Ε, αναφέρομαι και σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό Ράινφερτ στο Στρασβούργο που ανέφερε ακριβώς αυτό που είπα κατά λέξη και να συνδέσουμε ε, δημοσιονομικές υπηρεσίες και τραπεζικές υπηρεσίες περισσότερο με την πραγματική οικονομία. Δεν θεωρεί η Σουηδική Προεδρία ότι ήγηκε και η ώρα να κάνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Σουηδικής Προεδρίας. Σπέβδω να πω ότι θα φύγω πιο ευχαριστημένος από τη σημερινή συνεδρίαση, αν προλάβουμε, άλαβα απαντήσει σε δύο ερωτήματα. Κύριε Μπόργκ, είμαι από την Ελλάδα και την ώρα που μιλάμε τώρα κυριολεκτικώς πιθανόν να έχουμε προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών με αφορμή την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχει η χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση, συντηρητική κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζω, επανέλαβε και σήμερα το αίτημα να πάρει παράταση για τη μείωση των ελλημάτων. Απαντήστε μου λοιπόν, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Στο σημερινό ΕΚΟΦΗΝ συζητήθηκε το ελληνικό αίτημα. Έγινε δεκτό. Και γενικότερα ποια είναι η άποψή σας για τη γενίκευση αυτού του μέτρου, δηλαδή παράταση του χρονοδιαγράμματος για τη μείωση των ελλημάτων, σε χώρες που έχουν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που έχουν υψηλή ανεργία. Και ένα δεύτερο να σας πω πώς κερδίζουν οι ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα και να μου πείτε ε, τι μπορεί να γίνει. Το ελληνικό δημόσιο για να καλύψει τις ανάγκες εξέδωσε ομόλογα με επιτόκιο 5%. Τα ομόλογα αυτά τα αγόρασαν οι ιδιωτικές τράπεζες, τα εφάνισαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εγγύηση και πήραν δάνειο με επιτόκιο 1%. Τα κεφάλαια αυτά τα δίνουν σε επιχειρήσει, σε κτλ. και κερδίζουν με επιτόκιο 18% απομιζώντας, αν έγινε κατανοητό, τεράστια κέρδη χωρί κανένα κίνδυνο. Η ερώτηση λοιπόν κύριε Μπόργκ, δεν μπορεί να βρεθεί ένα άλλο τρόπο άμεση χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών των χωρών μελών παραδείγματο χάρη δανειοδότηση απευθεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μην επιτρέπουμε να λειτουργεί αυτό ο κερδοσκοπικό μηχανισμό. Σα ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τη Σουηδική Προεδρία. Αναφέρατε ότι μία από τις προτεραιότητες πρόκειται να είναι η ανεργία ή μάλιστα η απασχόληση. Αναφέρετε τα θέματα εργασιακής αγοράς. Θεωρώ ότι οι πιο ευέλικτες αγορές θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε τέτοιες συμφωνίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο ευέλικτες αγορές εργασίας. Θα πρέπει να είμαστε να αντιληφθούμε ότι το εργασιακό δίκαιο αποτελεί αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αναφορικά με τις προτάσεις και τις προτεραιότητες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Οι διερμηνείς θα μείνουν μαζί μας για 10 ακόμη λεπτά μάλλον 10 λεπτά επιπλέον, άρα έχουμε 7 λεπτά για τις απαντήσεις. Ευχαριστεί ευγενικά η Πρόεδρος τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος και ο συνάδελφός μου, ο κ. Ροντέλ, θα συμπληρώσει κάποιες από τις απαντήσεις που θα σας δώσω. για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και κατά πόσον θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ανάπτυξης, ελλείμματος, εκ παραλίλου. Θα πρέπει νομίζω να τονίσουμε, να υπογραμμίσουμε ότι αρκετές χώρες με υψηλό βαθμό απασχόλησης, όπως η Σουηδία, όπως η Δανία και η Ολλανδία, δεν ε, υπήρξε ε, επιδείνωση μεγάλη των δημοσίου χρέους. Άρα το δημόσιο χρέος δεν είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς την απασχόληση. Να πω επίσης ότι μπορεί να μην είσαστε ευχαριστημένος, αλλά φύγατε από το Συμβούλιο που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και πραγματικά εκτιμούσα ιδιαίτερα την περίοδο αυτή και τη συνεργασία μας. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την αγαστή συνεργασία υπό άλλους, ε, σε άλλες θέσεις πλέον. πλέον. Πιστεύω ότι η πρόβλεψη είναι ότι θα, θα καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία ε, για σημαντικά θέματα στο G20 και νομίζω ότι σημειώσαμε πρόοδο σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Ο κύριος Χόικμαρ έθιξε το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση. Δεν νομίζω ότι πολλοί καταλαβαίνουν την απάντηση. Δηλαδή ότι η ανάπτυξη του μοδησιοοικονομικού τομέα θα είναι πιο ε, εύστοχοι Το να μην δημιουργηθούν δηλαδή οι φούσκες που, που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε ε, δυνατά δημοσιονομικά πλαίσια και χρειαζόμαστε και πιο ευέλικτες αγορές εργασίας, πιο δυναμικές οικονομίες. Αυτή είναι η γενική απάντηση, αλλά νομίζω ότι με συγκεκριμένους όρους θα είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά την ανεργία Προφανώς υπάρχουν ε, κάποια σημάδια ανάκαμψης σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες, για παράδειγμα, των επιχειρήσεων. Αλλά η Ευρώπη παραμένει Ευρώπη. Ενώ η Άνοιξη μπορεί να έχει έρθει στο Νότο, στη Στοχόλμη έχει ακόμα χιόνι. Έχει ακόμα χειμώνα. Υπάρχει λοιπόν ε, και αυτό το στοιχείο. Έχουμε χειμώνα σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Υπάρχει απεσιοδοξία θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες για μεγάλη περίοδο ακόμα. Θα τηρήσουμε επιφυλακτική στάση και θα προσέξουμε την εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά την άμεση χρηματοδότηση του δημοσίου, των δημοσίων δαπανών από την ΕΚΤ, νομίζω ότι ενώ υπάρχουν πολλά προβλήματα στις αγορές, υπάρχει και μεγάλο στοιχείο πειθαρχίας και είδαμε ότι κάποιες χώρες Αυτό το σύστημα των ομολόγων αποτελεί ένα εγγενές στοιχείο της κρίσης, αλλά υπάρχει και ένα μακροπρόθεσμο στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία στον τομέα αυτόν. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάποια σχέση μεταξύ των στοιχείων αυτών. Το τελευταίο ερώτημα για το τι μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα για να βελτιώσουμε τις ε, αγορές. Οι πιο πολλές πολιτικές που σχετίζονται με την φύλαξη των παιδιών, με την εκπαίδευση, με τη βελτίωση των επαγγελματικών κινήτρων είναι σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να είναι σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία κοινοτική προσέγγιση. Αλλά τα βασικά θέματα, η εκπαίδευση, η φύλαξη των παιδιών, η φορολογία, η έρευνα, η ανάπτυξη, η κοινωνική ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Άντερς έδωσε ολοκληρωμένε απαντήσεις, οπότε εγώ απλά θα περιοριστώ το να πω ότι ήταν χαρά μου που παρευρέθηκα σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνατε για πολύ καλή συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και αναμένουμε να σας ξαναδούμε στο τέλος της Προεδρίας. Υπάρχει ένα σημείο στην ημερησία διάταξη. Να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 28 και 29 Σεπτεμβρίου.